of the agenda of today. And after... Και μετά από, αυτό, από αυτή τη γενική δήλωση της Επιτροπής θα στραφούμε στον αναφέροντα και στους συναδέλφους και ο κάθε συνάδελφος παρακαλώ σύντομα να παρέμβει. Λειτουργεί. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ε, δήλωση της Επιτροπής για τα ισπανικά υδρολογικά σχέδια από τον Μάρτιο. Αυτή η αξιολόγηση περιλαμβάνει πολλές σημαντικές πτυχές για τις αναφορές που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την συνεδρίαση. Και θα τα ακούσουμε και στις ερχόμενες παρεμβάσεις. Η Ισπανία συγκεντρώνει ένα σημαντικό ποσοστό της ε, εφαρμογής της οδηγίας για το νερό. Καταδικάστηκε το 2012 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ισπανία που δεν είχε κρίνει τα υδρολογικά σχέδια για όλες τις ε, λεκάνες απορροής. Ισχύει και πρέπει να γνωρίσουμε ότι έκαναν προσπάθεια τα τελευταία χρόνια οι Ισπανικές αρχές για τα σημαντικότερα επιρροτικά υδρολογικά σχέδια τα οποία εγκρίθηκαν το 2013 και το 2014. Αυτό το οποίο σημαίνει βέβαια σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με την προθεσμία του 2009 που προβλεπόταν στην οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι θα ανακτηθεί αυτή η καθυστέρηση και η πρώτη επικαιροποίηση θα γίνει το Δεκέμβριο του 2015 όπως προβλέπει η Οδηγία Πλαίσιο για τα Είδατε. αυτή την έννοια είναι θετικό το ότι οι δημόσιες διαβουλεύσεις για τα υδρολογικά αυτά σχέδια ξεκίνησαν το Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του Ιουνίου. Έχουμε εξαιρέσεις για τα Κανάρια που έχουν εγκρίνει όλα τα υδρολογικά σχέδια. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση, ε, στα Κανάρια παραλαμβάνω, και ελπίζουμε ότι θα λυθεί το ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Αναγνωρίζουμε ότι έγιναν σημαντικές τεχνικές προσπάθειες ε, για την κατάρτιση των Ισπανικών υδρολογικών Σχεδίων, ωστόσο αναγνωρίζουμε ορισμένα κενά στην εφαρμογή και έχουμε καταθέσει συστάσεις για βελτίωση της κατάστασης και συνοπτικά θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τα κενά αυτά στην εφαρμογή και τι σχετικέ μα συστάσει. Ο σημαντικότερο στόχο τη οδηγία πλαισίου για τα ύδατα είναι να αποτροπεί η επιδείνωση και να βελτιωθεί η κατάσταση των υδάτων. Εν γέννη τα υδρολογικά σχέδια δεν προσδιορίζουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποκατασταθεί καλή κατάσταση των υδάτων. Υπάρχουν πολλέ εξαιρεσει προ το στόχο αυτό και δεν δικαιολογούνται επαρκώ στα σχέδια η αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων δεν είναι πλήρης. Λείπουν οι μέθοδοι για την εφαρμογή των μέτρων και σε συγκεκριμένους ε, υδροφόρους όρους δεν έχουμε στοιχεία για το τι κατάσταση έχουν. Το κράτος δεν παρακολούθησε με επαρκή τρόπο την κατάσταση. Ουσιαστικά σε κάποιες λικάνες απορροής εγκατέλειψε τελείως την παρακολούθηση κατάστασης των υδάτων, όμως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, γιατί αν δεν γνωρίζουμε τι κατάσταση έχουν τα έδατα, δεν είναι δυνατό να γίνει η ε, διαχείριση του πόρου αυτού, του νερού δηλαδή, με το σωστό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ε, Ισπανία να ολοκληρώσει το μητρό υδάτων το στομότερο δυνατό, να κάνει την απογραφή, να υπάρχει έγκριση λοιπόν και καταγραφή θα πρέπει να γίνει και μία αναθεώρηση ώστε τα εξαγόμενα ύδατα να επιτυγχάνουν την αποκατάσταση της καλής κατάστασης των υδάτων λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους σπόρους. Θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να γίνονται μετρήσεις, έλεγχοι από πλευράς των αρμόδιων για τις λεκάνες απορροής αρχών και γι' αυτό κατεπηγόντως θα πρέπει να γενικευθεί η χρήση συγκεκριμένων μετρητών για την υδρολογική ροή και για να υπάρξει και καλή ποσοτική διαχείριση του πόρου. Σε σχέση με τη μέτρηση λοιπόν του ρυθμού της ροής και για την ανάκτηση του κόστους, έχουμε και τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για τα ύδατα, θα πρέπει να υπάρξει ένας ογκομετρικός συντελεστής για την ανάκτηση του περιβαλλοντικού κόστους από όλες τις χρήσεις του νερού και από τη χρήση των υπόγειων υδάτων. να συντελεστεί αυτό, αυτός όπως θα πρέπει να δώσει κίνητρα για την πιο αποτελεσματική χρήση του πόρου αυτού, όπως απαιτείται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Και έτσι θα επιτευχθούν και οι στόχοι τη εν λόγω Οι νέες υποδομές που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο ε, τους όγκους του νερού, όπω είναι τα μεγάλα φράγματα για παράδειγμα, θα πρέπει να αιτιολογούνται μόνο με βάση όρους που ορίζονται στο, στην οδηγία πλαίσιο. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ που να είναι και βιώσιμες και καλύτερες από περιβαλλοντικής πλευράς. Επίσης θα πρέπει να έχουμε οικολογικές ταχύτητες ροής για την καλή κατάσταση των υδάτων όπως είπα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, και οι προστατευόμενες περιοχές που εξαρτώνται από το νερό. Όταν καθορίζονται δηλαδή αυτές οι ροέ, ε, ροές, ε, υδρολικές ροές, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες των προστατευόμενων περιοχών. Σίγουρα όλα αυτά απαιτούν μέτρα πολύπλοκα από τεχνικής πλευράς. Τώρα, ε, δεν υπάρχει επαρκής ε, εφαρμογή των στόχων και των ε, μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία τα ύδατα σε ό,τι αφορά τα υδρολικά σχέδια της Ισπανίας, εστιάζουν σε δύο διαφορετικούς άξονες αυτά τα υδρολικά σχέδια. Πρώτος, παραδοσιακούς στόχους, δηλαδή ποσοτική διαχείριση του νερού και ανάπτυξη υποδομών για την ε, πλήρωση της ζήτησης, για την ικανοποίηση της ζήτησης και ο δεύτερος άξονας είναι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα που προβλέπει κάποια μέτρα, οικολογική κατάσταση, μέτρα για την ε, επίτευξη του στόχου της καλής κατάστασης ε, των όγκων νερού. Δύο διαφορετικοί άξονες λοιπόν που δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη και πολλές φορές είναι και ο ένας έρχεται σε αντίθεση με τον άλλον. θα πρέπει ε, να μην αυξηθεί με τις αρδευόμενες εκτάσεις η πίεση ε, στους, ε, στον υδροφόρο ορίζοντα. Το αντίθετο θα πρέπει να συμβεί. Τώρα η οδηγία πλαίσια για τα ύδατα παρέχει μια δυνατότητα πολύ σημαντική για την εκπλήρωση των στόχων μεν της οικονομικής ανάπτυξης αλλά χωρίς να βλαφθεί το περιβάλλον δε. Πρέπει να διατηρηθεί η ζήτηση. Έχουμε υπόψη μας και ότι μειώνονται ε, το νερό, δηλαδή λόγω των ε, αλλαγών στο κλίμα. Όλα αυτά καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία μιας πολιτικής που θα βασίζεται στις αρχές της αηφορίας, όπως προβλέπει και οδηγία πλαίσιο. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι Ισπανικές Αρχές προβαίνουν του τελευταίους μήνες σε μια διαρκή ανταλλαγή απόψεων. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν αναλύει τι απαντήσει των Ισπανικών αρχών στις δράσεις οποίες προτείναμε για τη βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας. Και αυτό σε σχέση με την έγκριση των δεύτερων υδρολικών σχεδίων στο τέλη του έτους 2015. Αν δεν θεωρηθεί απαρκής η πρόοδος και αν δεν υπάρξει μια αξιόπιστη δέσμες από πλευρά των ε, Ισπανικών αρχών για να διορθωθούν οι αδυναμίες, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί σωστά η οδηγία πλαισιοκοιτέρατα από την Ισπανία. Ολοκληρώνοντα αυτή τη γενική εισαγωγή, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εντοπίσαμε ότι πολλά τα προβλήματα που θα συζητηθούν σήμερα στο πέστον αναφορά είναι συστημικού χαρακτήρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι καλό θα ήταν τις καταγγελίες και τους ισχυρισμού των αναφερόντων να τις εξετάσετε με βάση και ε, τα ε, οριζόντια μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση των υδάτων με βάση τους όρους της οδηγίας πλησίου για τα ύδατα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα με οριζόντιο τρόπο εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την αποτελεσματική χρήση των πόρων και συγκεκριμένα του πόρου αυτού, του νερού δηλαδή, και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτό σε ό,τι αφορά ε, τη γενική μου τοποθέτηση και όταν μου δώσετε το λόγο θα σας ε, σχολιάσω την αναφορά που είναι στο σημείο 5 της Μερικής Διάταξης. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να τονίσω ότι σήμερα Θέλουμε οριζοντίω να δούμε όλε αυτέ τι αναφορέ μαζί, επειδή αυτό έχει και μια παιδαγωγική αξία για μας. Ακαδημαϊκή θα έλεγα, να τα καταλάβουμε σε περισσότερο βάθος και να τα δούμε ε, ενιαία στην σημερινή περίσταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτή τη γενική δήλωση για την όλη κατάσταση και θα επανέλθουμε ευθύς αμέσως σε εσάς. Και τώρα ο λόγος ε, στον κύριο ε, Σάντσεφ Πέρες, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την ε, πλατφόρμα στον ποταμό Τάγο και θα ξεκινήσετε με μια παρουσίαση PowerPoint, από ό,τι κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ναι. Έχω 30 διαφάνειες περίπου σε ένα PowerPoint για να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ποταμός ε, Τάγος, ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιβηρικής Χερσονήσου που διαβρέχει και την ε, Ισπανία και την ε, Πορτογαλία. Δεν είναι πριν από δεκαετίες αυτές οι φωτογραφίες, αλλά πολλές πριν από 5 ή 10 μέρες τραβήχτηκαν τον τελευταίο χρόνο τέλο πάντων περισσότερες Βλέπετε λοιπόν εδώ ε, την αναφορά μας ήδη από το 11 την καταθέσαμε η πλατφόρμα για την προστασία αυτών των ποταμών μαζί με την Καστίγια Λαμάντσα τα τελευταία χρόνια τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από 100 ενώσεις από την Ισπανία και από την Πορτογαλία συμπαρατάσσονται με την προσπάθειά μας και μιλώ και για την εκ μέρους μεγαλύτερη δήμου της ε, περιοχής μας. Δεν είναι ένα θέμα που θα το χαρακτηρίζει κανείς ε, δευτερεύον. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό που ίσως και να υπερβαίνει τα σύνορα και τα όρια της ε, του υδρολογικού σχεδιασμού στην Ισπανία ή της προσαρμογής ε, των υδρολικών σχεδίων όπως ε, ζητείτε στην οδηγία πλαίσιο. Τέταρτη φορά παρεμβαίνω στην Επιτροπή Αναφορών. Θα ήθελα να σας πω ότι τις τελευταίες φορές ε, ουσιαστικά αυτό που σας ζητούσαμε ήταν βοήθεια. Όμως ουσιαστικά δεν έχουμε πλέον χρόνο, δεν μπορούμε να στήσουμε πλέον βοήθεια, αλλά ζητούμε να δικαιωθούμε, δικαιοσύνη ζητάμε. Θα δείτε όσο μιλώ εγώ αυτές τις φωτογραφίες, βλέποντας αυτόν τον ποταμό, Βλέπετε την παραλία στο Τολέδο εδώ. Καμία σχέση δεν έχει με αυτό που είδατε πριν. Πάντα για το Τολέδο πρόκειται ή με αυτή την ε, φωτογραφία που βλέπετε τώρα του Τολέδο πάλι πριν από δύο χρόνια περίπου. Βλέπετε την υφή του νερού, την ποιότητα του νερού. Πολύ ξεκάθαρα πρέπει να σας πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Η Ισπανική κυβέρνηση εδώ έχει καταθέσει κάποια υδρολικά σχέδια για τον Τάγο και άλλοι θα σας μιλήσουν για άλλες λεκάνες απορροής, όλα φαίνονται θαυμάσια, καταπληκτικά. Και παρότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, μας τα είπε και ο κύριος Ροντρίγε Ρομέρο, φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια για την ε, διόρθωση κατάσταση. Δεν ισχύει αυτό όμω, στην περίπτωση του Τάγου στην Ισπανία, όπω είπα είναι ο μεγάλο ποταμό στην Ιβερική Χερσόνη, δεν είναι πλέον ποταμό, θα έλεγα, δεν λειτουργεί ω ποταμό, Είναι ένα οικοσύστημα που δεν λειτουργεί ως ποτάμι πλέον. Είναι μια σειρά από φράγματα ουσιαστικά και γύρω από το Τολέδο και άλλες πόλεις ε, ουσιαστικά είναι σαν ε, συλλεκτήρας ε, υδάτων, σαν μια λεκάνη συλλογής υδάτων. Και βέβαια χρησιμοποιείται για τη δόμηση, τη Μούρθια, τη Βαλένθια και για την άρδευση. Ε, στη, στην ακτή της Μεσογείου. Πριν από δέκα ημέρες ε, και για δύο εβδομάδες περίπου ο τάγος είχε μείνει για 80 χιλιόμετρα μήκος ε, στην κήτη του χωρίς νερό. Και όταν λέω χωρίς νερό, εμένα κάτι αυλάκια μόνο. Ήταν εντελώς στεγνός, στεγνή η κήτη του ποταμού. Έχουμε δει και στο Σανταρέμ στην Πορτογαλία κάποιες αντίστοιχες ε, εικόνες που βλέπετε ε, τι διαχείριση γίνεται στο ποταμό αυτό. Θα δείτε και πολύ άμμο εκεί. Ε, το θέμα είναι ότι θέλουν να υπάρξει μια εκτροπή το 80% του, των όγκων του νερού σε μια άλλη λεκάνη απορροής και εδώ βλέπετε κάποια ανάμιξη ε, υδάτων το 80% του καθαρού νερού με τα λίμματα. Υπάρχει, είναι αδύνατο να απορροφηθεί, να απορροφηθούν τα λίμματα τόσων εκατομμύριων ανθρώπων από αυτά τα καθαρά νερά. Επίσης έχουμε στην Εστρεμαδούρα ένα εργοστάσιο παραγωγής υδροελεκτρικής παραγωγής ενέργειας. και στην Πορτογαλία είχαν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα γιατί χρησιμοποιείται το νερό του ποταμού για αυτό το εργοστάσιο. Εδώ βλέπετε κάποια σε άλλες φωτογραφίες. Αυτή τραβήχτηκε στο Σανταρέμ πριν από λίγα χρόνια. Βλέπετε την άμμο που σας έλεγα γιατί είναι σχεδόν στεγνή κήτη του, του ποταμού. Καλό θα ήταν να έρθετε εκεί να δείτε πώς είναι ο ποταμός στην Ταλαβέρα, πώς είναι στο Τολέδο, πώς λειτουργεί η εκτροπή, για να δείτε ότι ουσιαστικά ε, στο σημείο από το οποίο πηγάζει ο ποταμός δεν υπάρχει νερό. 70% έχουμε ε, στη, στο σύνολο στην Ισπανία, στον υδροφορείο, 20-25% στις πηγές του τάγου. Υπάρχουν επίσης, ε, επίσης προστασίες κοινοτικού ενδιαφέροντος, υδρότοποι, ε, βιότοποι όπου κατοικούν ε, πτηνά, προστατευόμενες περιοχές, Natura 2000 και στον Τάγο υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που είναι τελείως αποξηραμένο νικήτη του ποταμού κινδυνεύουν και τα πτηνά. Γενικώ και η χλωρίδα και η πανίδα των προστατευόμενων αυτών κατά τα άλλα περιοχών Παναλαμβάνω λοιπόν ότι δραστικά κοροϊδεύει η Ισπανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον τρολογικό σχεδιασμό και προσπαθεί την τελευταία στιγμή να, κάνει, να, να πάρει κάποια μέτρα ή να καταρτήσει κάποια εντρολογικά σχέδια το οποίο είναι τελείως ε, αυτοσχεδιασμός και τελείως πρόχειρα σχέδια. πρέπει να ολοκληρώσω μάλιστα. Είναι ιδιωτική ε, ιδιοκτησία οι ε, ποταμή και οι εκβολές ε, και οι πηγές και για τη χρήση σε ηλεκτρικά εργοστάσια, όπως είπα. Αυτό το οποίο ζητούμε εμείς είναι η βοήθειά σας. Δεν μπορεί να στοιχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Πρόκειται για οικολογικό σκάνδαλο και για την Ισπανία και για την Πορτογαλία μιλάω. Κάποιο πρέπει να λάβει μέτρα. φαίνεται να κάνουν, να κάνουν ισπανικές αρχές ε, ε, καλά πράγματα, όμως ε, αν μας τραβήξουν λίγο τα αυτιά για τον τάγο και πάρουμε δύο-τρία λογικά μέτρα παραπάνω θα είναι όλα καλά. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν ε, κενά απλά στην εφαρμογή. Δεν εφαρμόστε καν αυτή η οδηγία πλαίσιο, κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν. Και ο καλύτερος μάρτυρας είναι οι φωτογραφίες που σας δείξαμε για το τι συμβαίνει. Σας ζητώ και ολοκληρώνω με αυτό να ληφθούν οι απαραίτητε δράσεις. Φυσικά ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Να έρθετε να δείτε το τάγο. Να μυρίσετε, να πιάσετε αν θέλετε και το νερό και να δείτε πώς γίνεται η διαχείριση αυτού του ποταμού. Στην Ευρώπη του 15, στην Ευρώπη του 16 πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ζητούμε από την Ευρώπη βοήθεια και κυρίως όπως είπα δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Η πρόεδρο σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα, για τη συγκεκριμένη αυτή αναφορά, επιστρέφω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αντιπροσωπευτικά τα ζητήματα της αναφοράς ε, σε σχέση και με όσα ανέφερα στην εισαγωγή μου, δηλαδή ότι πρέπει να εγγυηθούμε οικολογική, υδρολογική ροή, με στόχο, όπως είπα, και την αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων, ε, και να διατηρήσουμε και τις και περιστατευόμενες ε, περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από το νερό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με βάση αυτή την αναφορά προέδεισε ανταλλαγή απόψεων με, και πληροφοριών με την Ισπανική κυβέρνηση. πώς καταλάβαμε τα τελευταία στοιχεία, τα οποία και είμαστε στη φάση αξιολόγησης. Ε, αξιολογούμε αυτή τη στιγμή. Αναλύουμε κατά πόσον οι διαθέσιμες πληροφορίες αποδεικνύουν σημαντική επιδείνωση της κατάστασης διατήρησης ε, που οδηγεί σε καταστροφή ή υποβάθμιση οικοτόπων, οικοσυστημάτων και θέλουμε να δούμε και τη σχέση αιτίου και αιτιατού μεταξύ της ε, εκτροπής ε, του νερού και της υποβάθμισης ε, αυτών των πληγισσών προστατευόμενων περιοχών. Αυτά ευχαριστώ. Thank you very much. σας ευχαριστώ και εγώ. Ως γνωρίζετε, έχουμε ήδη αποφασίσει ότι θα διεξαράγουμε μια εξεταστική των πραγμάτων αποστολή για να δούμε τα πράγματα επιτόπου με τα μάτια μας. Νομίζω ότι μάλιστα σήμερα είναι και ιδιαίτερα επίκαιρη η περίσταση για να μπορέσουν τα μέλη μας να συλλέξουν τα απαραίτητες, απαραίτητες για να μπορέσουν να προχωρήσουν τη διεξαγωγή της αποστολής. Τώρα η κυρία Καμπεσόν έχει ζητήσει το λόγο και θα ακολουθήσει η κυρία Βαλίνα. Καλησπέρα σας. Αφού... Α, με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι εμένα δώσατε το λόγο, συγγνώμη. Συγγνώμη, Σολεδάτη. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, η σειρά δεν ε, είναι τόσο σημαντική. Αν ε, κατάλαβα καλά, θα συζητούσαμε από κοινού τι αναφορέ, γιατί ουσιαστικά εγώ έχω να κάνω και γενικά σχόλια για όλε αυτέ τι αναφορέ. Ε, ουσιαστικά το ίδιο θέμα είναι η ανάλυση των δρομικών σχεδίων και τι επιπτώσει έχει τελικά τη απορροή. Επομένως, ποια είναι η άποψή μου. Ουσιαστικά ε, μπορεί να υπάρξουν κάποιε διαφοροποιήσει ε, μικρέ ε, ανάλογα με την αναφορά, αλλά η θέση μου είναι η ίδια και είναι η εξή, ότι αφού ακούσουμε όχι μόνο τον πρώτο αναφέροντα, αλλά μάλλον αφού ακούσαμε και τον πρώτο αναφέροντα και την Κομισιόν και ήταν σαφή αυτά που είπαν, διαπιστώνεται δηλαδή ότι υπάρχουν κενά στα υδρολικά σχέδια που έχουν κατατεθεί και το θέμα αυτό το οποίο συζητούμε είναι πάρα πολύ λεπτό και βέστο. θα πρέπει να δώσουμε διεξοδικότατες απαντήσεις. Με βάση όλα αυτά λοιπόν πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε με αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτέ οι αναφορέ, να συνεχίσουμε ε, να συζητάμε το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την Επιτροπή Αναφορά αυτό το ζήτημα. Ε, Όμω ε, πραγματικά έρχονται εδώ οι αναφέροντε ε, και διαπιστώνουμε ότι ισχύουν αυτά που υποστηρίζουν τόσο καιρό. Πιστεύω λοιπόν ότι αξίζει να συνεχίσουμε να συζητούμε το θέμα αυτό, να μην κλείσουν αυτέ οι αναφορέ και κυρίω γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό λόγο συζητούμε για κάποια δραλογικά ε, σχέδια ε, τα οποία δεν ε, ουσιαστικά κυρώνονται διότι στα τέλη του 2015 υποτίθεται ότι πλέον πρέπει να υποβληθούν τα νέα, τα δεύτερα δραλογικά σχέδια. Δηλαδή έχουμε επιτάπτως κάποια δραλογικά σχέδια τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή παρουσιάσουν κενά σε σχέση με την οδηγία πλαίσια για τα ύδατα. Και από την άλλη πλευρά ακυρώνονται, καταργούνται αφού θα έχουμε τη δεύτερη γενιά δραλογικών σχεδίων. Νομίζω ότι το λογικό είναι να περιμένουμε τη υποβολή των νέων δρολικών σχεδίων, θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν διαπιστωθεί ότι αυτά τα κενά έχουν ε, συμπληρωθεί και καλυφθεί, μπορούμε ή δεν έχουν ανάλογα, θα πάρουμε μια σοβαρή απόφαση, όπως πάντα θέμα πολύ λεπτό, πολλά συμφέροντα, σύγκρουση συμφερόντων, ε, έντονα συναισθηματικά φορτισμένο το θέμα. Δεν ήταν σίγουρα σωστή η δεν εχουν αναλογα θα παρουμε μια σοβαρη αποφαση οπως το θεμα πολυ λεπτο πολλα συμφεροντα συγκρουση συμφεροντων εντονα συναισθηματικα φορτισμενο το θεμα δεν ηταν σιγουρα σωστη η καταρτιση των δρολικών σχεδίων. Αυτό είναι σαφές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα κυρία Βαλίνα. Τώρα Τώρα μάλιστα, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ε, όπως έλεγα και στην αρχή λοιπόν, αφού ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τους αναφέροντες, που δυστυχώς εντός εισαγωγικών, το λέω, γνωριζόμαστε από το 2012 ασχολούμαστε με αυτά τα προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση στην Ισπανία δεν έχει αλλάξει. Το αντίθετο ισχύει. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω το καθιστά απόλυτα σαφές. Και γι' αυτό επίσης ε, από τη δική μου πολιτική ομάδα επιμέναμε να ε, γίνει αυτή η επίσκεψη στον ΤΑΟ και στον Εύρο γιατί πρέπει να δούμε επιτόπου πώς έχει κατάσταση. Και φυσικά και πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά μέχρι ότου εκπονηθεί η έκθεση μετά την εκτασκευή των πραγμάτων αυτή επίσκεψη. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και την ε, Καλαβέρα εκεί, το σημείο που περνάει το ποτάμι και άλλα βέβαια σημεία. Είναι σημαντικό να επισκεφτούμε διάφορες ζώνες και του Έμπρο, όχι μόνο το Δέλτα, αλλά όταν περνάει και από τη Σαραγώσα, εκεί βλέπουμε στο σημείο αυτό να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Θα θέλαμε τώρα να υποβάλουμε μια πρόταση γενική. Όπως έλεγε η Σολεδάδ, ε, έχουμε να συζητήσουμε για ποτάμια από τη χώρα μας σήμερα, στο πίσω πολλών αναφόρων. Σε κάποιο κοντινό μέλλον και αν η κυβέρνηση δεν, πληρεί, δεν είναι ε, που λήγουν φέτος, στο τέλος της χρονιά, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο επιβολή κυρώσεων. Και αν πράγματι υποβληθούν αυτές οι ποινέ, αυτά τα πρόσφατα που θα πρέπει να πληρώσει η πανική κυβέρνηση θα πρέπει ε, να δοθούν ε, αυτά τα χρήματα, να δοθούν για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Για να τηρηθούν οι υποχρεώσει που έχει η χώρα μα ε, στο πλαίσιο αυτή τη οδηγία για, πλαίσια για τα υδατική επιτροπή αναφορών. Καλά ήταν να φτύνει μια επιστολή που δείχνει το ενδιαφέρον και την ε, ανησυχία μα για την κατάσταση των αναφορών και για τη συνέχεια που δίνεται σε αυτέ. Να στείλουμε σε όλε τι αυτόνομε περιφέρειε ε, και αυτόνομε κυβερνήσει αυτή την επιστολή. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Διώσο. Και θα ακολουθήσει η Μπεατρίση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θεωρώ ότι καλό είναι να τα συστήσουμε όλα από κοινού, αφού υπάρχει ένα κοινό παρονόμαστη που είναι αυτή η καθυστέρηση στην εφαρμογή τη οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα από την Ισπανία. Με βάση αυτή την οδηγία, το 2009 έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί τα υδρολογικά σχέδια για τι λεκάνε Το 2009 δεν υπήρχε κανένα ολοκληρωμένο υδρολογικό σχέδιο. Ξεκίνησε η κατάρτιση υδρολικών σχεδίων το Φεβρουάριο του 2012 μόλις. Άρχισαν τότε λοιπόν ε, να καταρτίζονται. Σήμερα έχουν υποβληθεί σχεδόν όλα. Ο πρώτος κύκλος δηλαδή των υδρολικών ε, σχεδίων. Η Κομισιόν έκανε τις παρατηρήσεις της, οι οποίες ε, θα ενσωματωθούν στο δεύτερο κύκλο υδρολικών σχεδίων. επομένω το πρόβλημα είναι από παλιά και νομίζω ότι έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν θέλω να επεκταθώ ιδιαίτερα γιατί έπονται και άλλες αναφορές που τα ίδια θα λένε και αυτές. Εδώ το πρόβλημα τελικά ποιο είναι. Έχουμε καθυστέρηση στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Μέχρι το 2011 δεν είχε ξεκινήσει να γίνεται τίποτα, απολύτως τίποτα. Άρχισαν ε, επί του τότε Υπουργού Άρια Κανιέτε ε, και είναι επιτρόπου να γίνονται κάποιες ε, προσπάθειε άρχισαν να καταρτίζονται τα υδραυλικά σχέδια. Και στα τέλη του 2015, έτσι προβλέπεται, πρέπει να χρονοκαθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναφορά αυτή, λέει ότι δεν υπάρχει καλή διατήρηση τη λεκάνη απορρίψη του τάγου, ιδίω μεταξύ ε, του, μέχρι το Καλαβέντελα Ρέινα και αναφέρει διάφορα στοιχεία λέει ότι δεν ε, γίνεται παρκή ζωολογικός καθαρισμός των λιμάτων όλα αυτά σίγουρα οφείλονται στην καθυστέρηση του σχεδιασμού, του σχεδιασμού επί της όμω όμως κυβέρνησης, σοσιαλιστική κυβέρνηση, το θέμα του 2011 δεν είχαν όπω όπως είπατε υδραλογικά σχέδια ούτε για τον τάγο επομένω. Άρα δεν ήταν δυνατόν το 2011 να έχουν επιληθεί αυτά τα προβλήματα. Το νέο υδρολογικό σχέδιο για τον τάγο εγκρίθηκε το 2014, πέρυσι δηλαδή, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το αξιολογήσει όπω και αν έχει εφαρμόσει τα νέα μέτρα ε, η Ισπανία, τα εντάσσει όλα τα υδρολογικά σχέδια του δεύτερου κύκλου σχεδιασμού. Και περί αυτού πρόκειται. Όλες αυτές οι αναφορές είναι πλέον ξεπερασμένες, αν θέλετε. Ε, είναι αναχρονιστικές. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεθέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Επιτροπής για όσα είπε που ήταν τόσο σαφή και ενδελεχή. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω στη συνέχεια των όσων αναφέρουν από τους αναφέροντες είναι το ότι εδώ είναι το σημείο κλειδί. Είναι θέμα και πρόβλημα συστημικού χαρακτήρα. Και σε αυτή την περίπτωση το θέμα δεν είναι το α, το β, η α, η β λύση. Αλλά το θέμα εντάξει έχουμε την οδηγία για τα ύδατα και έχουμε για τα πτηνά για τα προστατευμένα φυσικά περιβάλλοντα κλπ. Αλλά θα πρέπει να δούμε ολοκληρωμένα και να καταλάβουμε τι σημαίνει περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε καθυστέρηση τόσων ετών να μην τηρούνται οι υποχρεωτικοί κανόνες του κοινοτικού δικαίου. Ε, πρόκειται για θέματα ευρωπαϊκά και εθνικά. Μα είναι δυνατόν τα θεσμικά όργανα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να μην ε, υποχρεώνει προσημόρφωση είτε το κράτος ε, και να εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις να έχουμε αναμονή ενός, δυο και τριών ετών χιλιάδων ημερών ούτω ώστε να μπορέσουμε και να προσπαθήσουμε να άρουμε κάποιες ε, ανέκλητες ζημίες. Μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο γίνεται σε πολλά σημεία στην Ισπανία. Πρόκειται για το ότι θα πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτό το κοινό αγαθό η, η η ενιαία διαχείριση θα πρέπει να κατησχίσει. Και εμείς, επομένως προτείνω να αφήσουμε ως Επιτροπή ανοιχτές τις αναφορές, να ε, ενημερωθούν τα στοιχεία που έχουμε, να βρούμε τα στοιχεία που λείπουν και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε μια κρίση πλήρη και αντικειμενική. Δεν είναι δυνατόν για κάποια θέματα να περιμένει τόσα χρόνια. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανακτηθεί. Πώς είναι δυνατόν εκ των υστέρων να προσπαθούμε να επαναφέρουμε τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση. Πρόκειται για βασικά δικαιώματα και η μεταβλητή πιο σημαντική εδώ είναι ο χρόνος όπως και σε άλλες περιπτώσεις και εδώ νομίζω ότι το βασικό είναι ο ρόλος μας ως φωνή των Ευρωπαίων να ζητήσουμε εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και να πετύσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει όπως οφείλει να ενεργήσει και να ζητήσει την τήρηση των συμπεφωνημένων. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Όλοι σχεδόν μέχρι τώρα οι Ισπανοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο και να είστε βέβαιες και βέβαιοι ότι θα αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε όλες αυτές τις διαφορετικές αναφορές. Όπως είπατε και εσείς κύριε Αγιούσο και άλλοι, υπάρχει όντως μια γενική προσέγγιση, δομικά δηλαδή προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μια αναφορά ξεχωριστά σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς. για να δουν και οι αναφερόμενοι, είτε βρίσκονται στην πατρίδα τους, είτε βρίσκονται εδώ, ότι όντω η αναφορά τους βρίσκει απήχηση στην Επιτροπή Αναφορών. Δεν είναι αναγκαίο να λάβετε το λόγο για αυτές τι αναφορέ που μιλήσαμε μέχρι τώρα, έρχονται και άλλε. μακρός κατάλογος. Άρα προσπαθήστε να αυτοπεριοριστείτε λίγο. Θα ακολουθήσει ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είναι σύντομο. Και Όπω είπα στην προηγούμενη συνεδρία, θέλω να σας πω ότι είμαι από εκεί. Ζω κοντά στι όχθε του Τάγου. Και θα πούμε τι γίνεται με αυτά τα προγράμματα για την ε, φυσική αυτή λεκάνη, τι γίνεται γιατί το θέμα είναι κατά πόσον τα όσα λέει η οδηγία αντιστοιχούν αυτό το οποίο γίνεται για την ποιότητα των υδάτων, για την ποσότητα των υδάτων επίσης. Οπότε το πρόβλημα είναι διτό, ποσότητα και ποιότητα. Οπότε και αυτά τα δύο προβλήματα δεν επιλύονται σίγουρα με αυτό το πρόγραμμα της Λεκάνης σε σχέση με τις δημοτικές αρχές ε, ε, πέραν των πολιτικών παρατάξεων. Όλοι, όλοι, από όλο το πολιτικό φάσμα είναι κατά Ούτε έγινε καμία ζήμωση, κανένα διάλογο. Εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή των ε, Αναφορών θα πρέπει να αξιολογήσει ό,τι γίνεται με αυτά τα ποτάμια. Αλλά θα πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα και θα πρέπει να δούμε πώ θα τελειώσουν να συμμεθούν τα κράτη-μέλη. Γιατί η... η στάθμη των υδάτων ήταν κοντά στο μηδέν ενώ θα πρέπει να είναι 10. Τέλος πάντων η ροή 10 ανά δευτερόλεπτο στα διάφορα σχετικά σημεία. Αλλά είμαστε πολύ παρακάτω από το κατόφλι το οποίο ε, θα πρέπει να ισχύει. Άρα δεν τηρούμε την ε, οδηγία. Αυτό το πρόγραμμα της λεκάνης δεν τηρεί ούτε κατά την ποιότητα ούτε κατά την ποσότητα. Είναι λανθασμένες οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Άρα θα πρέπει να εγγυηθούμε τη λήψη των αποφάσεων ως Επιτροπή Αναφορών και ως Κομισιόν Πρόεδρος. Το έχουμε ακούσει μέχρι τώρα πέντε σπανούς ε, συναδέλφους και ήρθε τώρα η ώρα για την Ιταλίδα συναδέλφο. Κυρία Εύη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ, και εγώ νιώθω το ίδιο αποτεμένο όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοι Πώς να μην συμφωνήσω. Βεβαίω και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον αγώνα που δίνουν οι αναφερόμενοι τόσα χρόνια. Γιατί πρόκειται για πολλά χρόνια που κουβεντιάζουμε τα ίδια, αναφέρονται τα ίδια για τα ίδια θέματα και λύση δεν βρίσκεται. Και όλα αυτά τα οποία τώρα ακούσαμε είναι η ουσία του προβλήματος. Η ποσότητα και η ποιότητα των υδάτων. Και οι δύο αυτές ε, μεταβλητές βρίσκονται αυτή τη στιγμή μακράν των όσων ορίζει ως στόχο ε, η οδηγία για να έχουμε ύδατα όπως πρέπει να είναι και να ε, υπάρχουν εγγύησεις ανάπτυξης του οικοσυστήματος. Να μην έχουμε επιδείνωση των συνθηκών και καταστάσεων. Επομένως, είναι να καταλάβουμε πολύ βασικός πόρος φυσικός στο νερό. Άρα θα πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Αυτό είναι το Και είναι απαράδεκτες οι σχετικές καθυστερήσει. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ασκήσουμε πίεση, γιατί πρόκειται για κάποιες πολιτικές επιλογές που βρίσκονται πίσω από αυτή την κατάσταση. Και θα πρέπει αυτές οι επιλογές να αλλάξουν το συντομότερο. σε αυτό το επίπεδο έγινε κάποια διαβούλευση όπως παρουσιάστηκε ε, αλλού δεν έγιναν αυτές οι διαβουλεύσεις δεν μπόρεσαν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί οι πολίτες γιατί μόνο από τους πολίτες και τον έλεγχο που ασκούν μπορούμε να έχουμε την ε, ουσιαστική εφαρμογή αυτής της οδηγίας στην Ευρώπη. Άρα μόνο χάρη σε αυτούς που επί επιτόπου κάναν την εξακρίβωση των όσων γίνονται προχωρήσαμε. Θα πούμε για τι γενικέ επόμενε αναφορέ, αλλά σίγουρα και αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλώς όρισαν οι αναφερόμενοι. Θέλω να πω ότι ζητεί βοήθεια, ζητεί δικαιοσύνη και αυτό και θα γίνει εδώ, αλλά όμω δεν είναι σωστό να πούμε ότι μα εξαπατάει η κυβέρνηση. Ούτε είναι σωστό να λέμε ότι τίποτα δεν άλλαξε στην Ισπανία. Βεβαίω και κάτι άλλαξε. Το 2009 ήταν ο πρώτο κύκλο αυτών των προγραμμάτων. Δεν έγινε τότε τίποτα, γι' αυτό δικαστήκαμε και ορθώ. Τώρα όμω η κατάσταση είναι ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτο κύκλο, οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε ό,τι πρέπει να αλλάξουμε και αυτό που οποίο προβλέπεται είναι πριν το Δεκέμβριο του 2015 να έχει γίνει κάτι. Βεβαίω. Άρα κάτι άλλαξε. Ίσως τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο θα ήθελαν οι αναφερόμενοι και εμείς, αλλά κάτι έγινε. Τώρα για την Κομισιόν. Η έκθεσή σας ήταν πάρα πολύ αυστηρή και σκληρή. Ίσως ορθώς, αλλά δεν θα πρέπει να κολλάμε στο ιστορικό, στο παρελθόν, στο τι έπραξε η Ισπανία γιατί όπως είπαμε θα πρέπει να αξιολογηθεί το τι έκανε η Ισπανία. Αυτό θα πρέπει να διαπιστώσουμε. Προγραμματισμός, συζήτηση, ζήμωση και όχι εκθέσεις να βασίζεται στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη τα νέα προγράμματα, τις τροποποιήσεις οι οποίες προτάθηκαν. Και αυτή η έκθεση περισσότερο αφορά το παρελθόν παρά το παρόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Muchas gracias. Now, Senor Terry Cabras. Thank you, Chair. Since it has already been said... Επειδή λέχθηκε ήδη η άλλοι συνάδελφοι, δηλαδή όσα θα ήθελα να πω και είμαστε πέρ του αναφερομένου, ε, γι' αυτό και εγώ ε, θεωρώ ότι καλύφθηκα και δεν ε, θα μιλήσω. Ο κύριος Ουρτασούν. Κύριε Σαρταζούνη, θα είμαι σύντομο για να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ πέρα με τόση όρεξη για να καταγγείλουν αυτές τις κατάφορες παραδιάσεις της Ισπανίας για τα ύδατα. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτές οι αναφορές παραμένουν, παραμένουν επίκαιρες. Ε, είναι, είναι, είναι της καυτής επικαιρότητας και έχουμε αυτή τη σκληρή έκθεση της Επιτροπής η οποία αναφέρεται στα κενά που έχουν αυτά τα προγράμματα. Δεν είναι θέμα το ότι είναι κολλημένη στο παρελθόν η Κομισιόν. Αυτό έγινε και αυτό συζητάμε. Ήθελα να λάβω τον ε, λόγο νωρίτερα για να ζητήσω ότι θα πρέπει να μείνουν ανοιχτέ οι αναφορές όσο κάνει την αξιολόγηση των ε, προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως θα πρέπει να κάνουμε μια αποστολή επιτόπου. Το θέμα έχει τραβήξει πάρα πολύ και θα πρέπει και η Κομισιόν και η Επιτροπή των Αναφορών να πάρουν στα σοβαρά τα πράγματα. Άρα, το σωστό είναι, λέει η πολιτική μας ομάδα, να μην είναι ανοιχτή η αναφορά. Οι αναφορές. Και προτείνουμε επίσης να γίνει και αυτή η αποστολή επιτόπου. Νομίζω θα ήταν πολύ σωστό. Ακριβώς αυτό προτίθεται να πράξει η Επιτροπή Αναφορών. Τώρα, λοιπόν, θα επιστρέψω το λόγο στους αναφερομένους και θα κάνω και κάτι ασυνήθιστο. Θα προσκαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σύντομα στις ερωτήσεις που έκαναν ο κ. Σμάτο και άλλοι. Αλλά παρακαλώ, εσείς ε, με την αναφορά λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που βλέπετε και με τις διαφάνειες είναι το σήμερα είναι ότι τι γίνεται πριν από μια εβδομάδα. Άρα δεν μιλάμε για το παρελθόν, δεν μιλάμε για ιστορία. Για να απαντήσω στους κυρίους, ε, στην κυρία Γιούσο και στον κύριο Μάτο. Το πρόβλημα του τάγου δεν είναι θέμα καθυστέρηση, είναι δομικό το πρόβλημα. Το υδρολικό σχέδιο για τη λεκάνη του τάγου αντί να προσαρμόζει την κατάσταση της πανική νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και να προβαίνει σε μια διαχείριση του ποταμού με βάση προηγμένες ε, ευρωπαϊκές παραμέτρους, ε, αυτό που κάνει είναι ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο του παρελθόντος, δηλαδή ουσιαστικά τον καταδικάζει σε ε, ισόβια κάθριξη κατά κάποιο τρόπο. Ε, τον φυλακίζει τον ποταμό αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα η αναθεώρηση των υδρολικών σχεδίων. Το ξέρω κυρία Γιούσο, κύριε Μάτο, τα έχω μελετήσει, ξέρετε. Ε, δεν ξέρω αν είναι δυνατό, αλλά μακάρι να μίλαγα ε, με τον καθένα και την καθημεία από εσάς για να αναλύσουμε κάθε ώρα και κάθε σελίδα ε, τι, τι γίνεται και να δείτε τι είναι αυτή, ε, αυτά τα νέα Ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, φυλακίζεται ο τάγο ε, και καταδικάζεται σε ισόβιο κάθερξη με αυτά τα υδρολικά σχέδια μέχρι το 2020 τόσο. Οι φωτογραφίε που σα έδειξα είναι αποτέλεσμα ε, του υδρολογικού σχεδίου του 2014 για τον τάγο. Και για να ολοκληρώσω, επειδή δεν θέλω να ε, επεκταθώ, μία σκέψη μόνο. Αφού εγμέκρινε αυτά τα σχέδια για τι λεκάνε απορροέ στη νομοθεσία τη Ισπανία, τροποποίησε την νομοθεσία, δηλαδή σαν να μην έφτανε σαν να μην ήταν αρκετά αρνητική η νομοθεσία για τη διαχείριση του τάγου συγκεκριμένα, τι έκανε η Ισπανία. Τροποποίησε κάποια, μάλλον κάποια βασιλικά διατάγματα και συγκεκριμένα μνημόνια συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων αυτόνομων περιφερειών, συγκεκριμένων περιοχών, για να στρεβλώσει, αν μπορώ να το πω, και να στραγγαλίσει ακόμη περισσότερο το τάγο και να αφήσει τη στάθμη του τα κατώτερα επίπεδα. Και κάτι τελευταίο, ο Τάγος είναι ο μόνο από τα μας από όλους όσους διαβρέχουν την ειδική Χερσόνηση, για τον οποίο δεν υπάρχουν οικολογικέ ε, υδρολικές ροές στο μέσο τμήμα του, το ΜΕ, στο Τολέδο, τα Λαμέρα, τα κτλ. Μπορεί λοιπόν το κράτο όπω έκανε για το παρελθόν, όχι πριν από 2-3-5 χρόνια, πριν από 10 μέρε. Μπορεί λοιπόν το κράτο όπω έκανε λοιπόν και τον νέο να παραβιάζει ε, τι διατάξει ε, τη νομοθεσία. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε ότι θα αλλάξει κάτι με αυτά τα νέα υδρολικά σχέδια. Ουσιαστικά θα τον βάλουν στο κελί του πάλι τον τάγο και θα τον αφήσουν εκεί μέχρι να σαπίσει. Thank you. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ροδρίγε Ρομέρο, αν επιθυμείτε παρακαλώ να απαντήσετε, έχετε το λόγο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω. Θα απαντήσω σε δύο σημεία. Πρώτα-πρώτα για τον παράγοντα χρόνο. Δίνεται η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστέρησε και ότι είχε συμπεριφορά αμελή όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τα ύδατα, αλλά και άλλων οδηγιών που αφορούν το περιβάλλον. Φερρυπή, να επενθυμίσω ότι εμείς έχουμε εισαγάγει τέσσερις περιπτώσεις ε, παραβίας του κοινωνικού δίκαιου στην Ισπανία. Μιλάμε για εκατοντάδες ε, δήμων και κοινοτήτων στην Ισπανία. Και επίσης έχουμε ανοίξει κάποιες διαδικασίες που αφορά ε, την παράληψη σύνταξης προγραμμάτων διαχείρισης για προστατευμένες ζώνες. Άρα, λαμβάνουμε κάποια μέτρα ούτως ώστε η τρευματική νομοθεσία να εφαρμοστεί. Η δε οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ε, έχει υποστεί καθυστέρηση στην εφαρμογή της σημαντική. Οπότε απλώς προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται με αυτά τα υδρολογικά προγράμματα τα στα τέλη περασμένου έτους και είχαμε ε, δυναμική συνεργασία με τις Ισπανικές Αρχές. Ανταλλαγή πληροφοριών. Συνεχή. Και τώρα. Οπότε είμαι σε θέση να σας πω ότι όλα τα θέματα τα οποία εφήγησαν δεν θα λυθούν όλα στη δεύτερη φάση γιατί υπήρξε πάρα πολύ ε, μικρό διάμεσο διάστημα μεταξύ της πρώτης φάσης και της δεύτερης τώρα το 2015. Πάντως ελπίζουμε ότι θα έχουν κάποιο αξιόπιστο σχέδιο οι Ισπανικές Αρχές ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και έτσι το νωρίτερο δυνατόν ε, αυτές οι παραλήψεις θα αρθούν. Στις εβδομάδες θα έχουμε μια συγκέντρωση, μια συνεδρίαση που θα αφορά ακριβώς την κατάσταση της πολιτικής των εδάτων στην Ισπανία. Ε, θα υπάρξουν και κάποια νομοσχέδια σχέδια. Οπότε θεωρούμε ότι ελπίζουμε θα βελτιωθούν τα πράγματα και ότι θα έχουμε κάποια σχέδια και προγράμματα αξιόπιστα το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όντως μπορούμε να λάβουμε απόφαση τώρα ε, επί της αναφοράς αυτής. Εγώ θα προτείνω να διατηρηθεί βεβαίως η αναφορά ανοιχτή. Να, όπως σας εξήγησα πριν, να διεξαγάγουμε την αποστολή επιτόπου Ιανουάριο-Φεβρουάριο Φεβρουάριο του 2016 στην Ισπανία για να δούμε με τα μάτια μας την κατάσταση και για να προετοιμαστούμε για αυτή την αποστολή, την εξεταστική αποστολή να προσκαλέσουμε ενδεχομένω και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέλθει και να μας ενημερώσει για τα πιο πρόσφατα γεγονότα καθώς και εκτιμήσεις που θα έχουν γίνει ίσως μαζί και με εκπροσώπους των Ισπανικών Αρχών έτσι ώστε να είμαστε καλά προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι για την εξαγωγή της επιτόπου αποστολής. Εάν δεν υπάρχει οτιδήποτε επιθυμεί να μας υποβάλει γραπτός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα έχει νέες πληροφορίες. Το ίδιο ισχύει και για τις Ισπανικές Αρχές. Εφόσον έχετε νέες πληροφορίες που επιθυμείτε να τις θέσετε υπόψη της Επιτροπής Αναφορών, να το πράξετε και πολύ ευχαριστώ να δεχτούμε οποιασδήποτε νέες πληροφορίες μπορούμε να έχουμε από εσάς. Είστε σύμφωνες και σύμφωνοι? Ωραία λοιπόν. Τότε ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτού του θέματος. Και ως γενικό συμπέρασμα, ισχύει βέβαια για αυτή την αναφορά, αλλά και για τις άλλες που θα συζητήσουμε σήμερα, αυτό που θα πρέπει να πράξουμε όλες και όλοι μας, θα πρέπει να είναι να ε, εκμεταλλευόμαστε ορθά, λογικά την φύση, χωρίς να την υπερεκμεταλλευόμαστε και χωρίς να την καταστρέφουμε. Έχουμε τώρα την 0938 Ματίλντε Φοντέν της Κορδιναδόρα Αντιτρανσβασαμέντς για τον ε, Ισπανικό ποταμό Εύρο. Ισπανικό ποταμό Εύρο. Και είναι παρούσα η αναφερομένη. Ε, ο αναφερόμενος. Πολύ ευχαρίστως να σας δώσω τον λόγο Φοντ Τέν, έξω ονόματος της οργανώσεως που εκπροσωπείται. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, καλημέρα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή που έχει τύχει η υπόθεσή μα από τη πλευρά. Εμεί προερχόμαστε από το Δέλτα του Ποταμού Εύρω. κοινωνικό κίνημα ο οριζόντιου χαρακτήρα και εδώ και 30 χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε τις κατά καιρούς κυβερνήσεις της χώρας μας ότι ζούμε σε κάποιο χώρο μοναδικό, πάρα πολύ ευάλωτο και με οικολογική αξία. Ε, ζούμε στις εκβολές του Εύρου και ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ η διατήρηση να καθιστά ε, συμβατή τη χρήση για τη γεωργία και από πλευράς ε, αστικής χρήσης να είναι όλα αυτά όπως πρέπει για να προστατευτούν τα ύδατα του Δέλτα. Έχουμε 320 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκεί. Ε, είμαστε 60.000 κάτοικοι. Πρόκειται για το τρίτο πιο μεγάλο δέλτα της Μεσογείου μετά την γαλλική Καμάρντ και το δέλτα του Νείλου. Είναι πολύ σημαντική, σημαντικός υγροτόπος και εκεί έχουμε αποσπάσει κάθε διεθνή προστασία υπάρχει. Είναι ζώνη Ραμσάρ, Ζέπα, ΛΙΚ για το Natura 2000 και το 2013 ε, επίσης θεωρείται προστατευόμενη ζώνη της βιοσφαίρας. Στις 9 Εβδόμου του 2013 η πλατφόρμα προστασίας του Εύρου ε, προσέφυγε πρώτη φορά στην Επιτροπή σας. Τότε που η Ισπανική κυβέρνηση ε, κατέβασε αυτό το σχέδιο υδρολογικού προγράμματος και εκεί χωρίς να το δικαιολογεί έλεγε ότι θα ε, προβεί σε έργα ίδρευσης πάνω από 450.000 νεκταρίων και 40, και 40 ε, νέες τεχνητές λεκάνες υποδοχής υδάτων. Και είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία αυτού του οικοστήματος από το Ευρωπαϊκό Δεστός. Και ελπίζαμε ότι κάτι θα γίνει και να μην μας αφήσετε μόνοι μας. Στις 28 Δευτέρου του 2014 η κυβέρνηση της χώρας ενέκρινε χωρίς καμία τροποποίηση αυτό το υδρολογικό πρόγραμμα της λεκάνης του Εύρου, ακριβώς όπως είχαμε επισημάνει ενώπιν της Επιτροπής σας. Στις 19 Ενδεκάτου του 2014, μια από πια είχαμε ε, νόμο του κράτους που είχε εγκριθεί ε, να σε αυτήν την ένσταση ενώμης Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπαμε ότι έχει παραβιαστεί η οδηγία για τα άγουα, για το φυσικό περιβάλλον, το προστατευόμενο και για τα πτηνά του 2014 και είπαμε για δεύτερη φορά εδώ μπροστά ότι παρά το όσο πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, είδαμε καμία προσπάθεια πλευρά τη Ισπανική κυβέρνηση να υπάρξουν κάποιε ουσιαστικέ αλλαγέ σε αυτό το κείμενο του, του υδρολογικού προγράμματο για τον Εύρο, ούτε είχαν ληφθεί υπόψη οι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στι 13 Πέμπτου 2015 ε, ελάβαμε μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σύμφωνα με αυτή την επιστολή, το υδρολογικό σχέδιο ή πρόγραμμα του Εύρου βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης και δεσμεύτηκε η Ισπανική αναθεωρησης και δεσμευθηκε η ισπανικη κυβερνηση να λάβει υπόψη τι συστάσεις ή στην ε, περίοδο ε, ενό μηνό όμως η ένστασή μα μπήκε στο αρχείο. Εμεί έχουμε κάνει και άλλα διαδήματα και υποβάλαμε κάθε τεκμηρίωση ούτω ώστε να μην έχουμε αυτή την θέση στο αρχείο τη ενστάσεώς μα. Σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι η έγκριση του προγράμματο ε, για τον Σεπτέμβριο φέτος αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ουσιαστική τροποποίηση, του 500, τι θα γίνει με, αυτό, με αυτά τα με αυτά τα ποτιστικά σχέδια που υπάρχουν για αυτά τα 400.000 εκτάρια για τις 40 τεχνητές ε, λίμνες υποδοχής υδάτων για το δέλτα του Εύρου. Ούτε, ούτε εκεί θα υπάρξει καμία τροποποίηση και οπότε τώρα είπαμε ότι θα πρέπει να βρούμε ε, κάποιο είδους ε, βασικούς πόρους Και σας ευχαριστούμε κύριοι βουλευτές γιατί βοηθήσατε να κάνουμε αυτό το τρίτο διάφημα εμείς ως πλατφόρμα για την προστασία του εύρου και παρακαλώ μην μας εγκαταλείπετε και να μην κλείσετε την αναφορά. Πρόκειται για 60.000 ε, που ζούμε στο Δέλτα και ε, αισθανόμαστε απροστάτευτοι Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, ούτω ώστε να ζητηθεί από την κυβέρνηση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της σε σχέση με την Ένωση, αλλά και να εφαρμόσει την οδηγία για τα ύδατα. Παρακαλούμε εμποδίστε την κυβέρνηση να διασπαθίζει το δημόσιο χρήμα, ε, όπως επίσης και το χρήμα των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Δεν νομίζω ότι ζητούμε τίποτα το τρομερό, απλώς να τηρηθούν οι διατάξεις και κατευθύνσεις που ορίζουν ε, τα θεσμικά όργανα επίσης παρακαλούμε να στείλετε μια αντιπροσωπή της Επιτροπής σας στο ΔΕΛΑ του Εύρω και έτσι επιτόπου να εξετάσετε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του ιδρυολογικού προγράμματος για ε, την ε, λεκάνη του Εύρου όπως ενεκρίθη πέρσι. Τώρα θέλουν να κάνουν μια αναθεώρηση αλλά ουσιαστικά δεν αλλάζουν τίποτα και η οριστική έγκριση θα γίνει κατά τα τέλη του τρέχοντος έτους. Εν να σας πω ότι αυτό το οποίο θέλουμε εμείς από τη γη του Εύρου ε, είναι το να βελτιωθεί αυτό το πρόγραμμα, να προστατευθεί ε, το Δέλτα του Εύρου και ό,τι κάνετε θα μας βρει πάντα συμμάχους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και ιδιαίτερος για την υπομονή σας να προσέρθετε για τρίτη φορά στην Επιτροπή Αναφόρων. Ναι αποστολή που θα οργανώσουμε στις αρχές του επομένου έτους, ακόμα δεν έχουν οριστεί οι ημερομηνίε, αλλά θα περιλάβουμε και τον ποταμό Έμπρο ε, στο αντικείμενο που θα εξετάσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν για την υπομονή σας και θα ήθελα πάλι να σταθώ τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την, ειδική, για την συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Μας ε, είπατε την οριζόντια άποψή σα για τι διαστατικέ αυτέ μεταβολέ, αλλά είμαι βεβαία ότι και εδώ θα έχετε κάτι χρήσιμο να προσθέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτήν την αναφορά τα ζητήματα που θεωρούμε επίσης ότι είναι δομικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κακή εφαρμογή τη οδηγία πλαισίου για τα έδωτα από την Ισπανία δεν αξιολογήθηκε επαρκώς η κατάσταση των υδάτων και αυτό επηρεάζει σίγουρα και τα επόμενα στάδια του σχεδιασμού, διότι Εάν δεν είναι πλήρε το πρώτο στάδιο αυτό τη αξιολόγηση τη κατάσταση, όπω συμβαίνει στο Δέλτα του ΕΜΠΡΟ, δεν μπορούν να, να καταρτιστούν περιβαλλοντικοί στόχοι, άρα ούτε και τα κατάλληλα μέτρα μπορούν να θεσπιστούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Ισπανία έχει εργαστεί εντατικά, αναπτύσσει μεθόδους ε, για την δημιουργία υδρολογικών ε, ροών και σε εθνικό επίπεδο όμως αυτές οι υδρολογικές ροέ οι οικολογικές δεν συνδέονται ξεκάθαρα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της οδηγίας πλαισίου. Ούτε με τους στόχους για την προστασία των ε, περιοχών ε, που την χάνουν ε, προστασίες όπως είναι ή πρέπει να είναι το Δέλτα του Εύρου. Υπάρχουν διάφορα σχέδια υποδομών, περιλαμβάνονται και στο υδροϊκό σχέδιο για το Δέλτα του Έμπρο, φράγματα μικρότερα και μεγάλα που δεν έχουν δικαιολογηθεί, σύμφωνα τουλάχιστον με την οδηγία για τα ύδατα δεν δικαιολογούνται. Ε, πριν από λίγες εβδομάδες ξεκίνησε η διαδικασία του παραβάση κατά της Ισπανίας ε, σε ό,τι αφορά το φράγμα του Μπισκαρουές που βρίσκεται σε αυτή τη λεκάνη απορροής του Εύρω. Ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύει ότι το θέμα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη στο μελλοντικό υδρολογικό σχέδιο. Τώρα, όταν τα έργα αφορούν ε, όγκους νερού για τους οποίους δεν έχει εκτιμηθεί η κατάσταση και δεν έχουν ε, καταρτιστεί περιβαλλοντικοί στόχοι, πρόκειται εδώ για μια λεκάνη απορροής που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ε, υδάτων που δεν γνωρίζουμε τι κατάσταση, τι κατάσταση κολλική βρίσκεται. Υπάρχει κενό στην ενημέρωση. Πολύ δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί κανείς το πρόβλημα αυτό για να κάνω σωστό σχεδιασμό. Όπως προανέφερα, στην αρχή μου τουλάχιστον παρέμβαση είχα πει ότι συμπεριλάβαμε την εξέταση των καταγγελιών στις οριζόντιες δράσεις μας ε, για την βελτίωση της άμεσης οδηγίας και θέλω να διαβεβαιώσω και τους αναφέροντες και την Επιτροπή σας ότι το γεγονός ότι αυτή η καταγγελία ε, έχει υπάρξει πρόταση να αρχιοθετηθεί αυτό οφείλεται στην ε, αποτελεσματικότητα και διοικητική οικονομία εντό αγωγικών. Όχι δεν θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της απταγγελίας, θα ενταχθούν, όπως είπα, στις οριζόντιες μας δράσεις. Που έχουν αυτές οι δράσεις στόχο τη βελτίωση τη εφαρμογή οδηγία στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now the floor is open to members. First of all... Είναι ανοιχτό ε, ανοίγει τώρα η συζήτηση, μπορείτε να λάβετε το λόγο, τα μέλη και κύριε Μαρτάν πρώτος εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώντας τα όσα εξηγεί η αναφερομένη, θυμούμε άλλες παλαιότερες αναφορές, διότι η παρούσα αναφερομένη ε, και σε συνδυασμό και με την προηγούμενη για τον Τάχο, με ανησυχούν αυτά, διότι εάν πιστέψω τα όσα λέγονται, από 400.000 εκτάρια ε, έχει περιοριστεί πολύ και πρόκειται να ήδη να αρχίσει. Μα είπε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όντω και αυτό το επανέλαβε και η αναφερομένη, δεν έχουμε ακόμα επαρκείς εκτιμήσει σχετικά με τι ενδεχόμενε επιπτώσει του έργου. Η απάντησή μου λοιπόν είναι απλή. Εγώ επιθυμώ όντω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, επιθυμώ να γνωρίζω σοβαρά τις επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα και να προβεί σε διαβήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην Ισπανική κυβέρνηση για να ανασταλεί η εκτέλεση του έργου πριν να γνωρίζουμε πραγματικά ποιε θα είναι οι επιπτώσει. Ορίστε κυρία Πρόεδρε, αυτά πω. Η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούστε. Οι αναφέροντες αμφισβητούν την πρόταση υδρολικού σχεδίου για τον Εμπρο από το 2012 ότι παραβιάζει πολλές οδηγίες. Η πλατφόρμα αυτή τη θέλει όμω ουσιαστικά αυτή η οικολογική υδρολική ροή ε, που έχει φτάσει, ε, θέλει να φτάσει σε τριπλασιασμό ουσιαστικά ε, του όγκου του νερού. Αυτό το υδρολικό σχέδιο για τον Εύρο όμως εγκρίθηκε το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μελέτησε. Στο δεύτερο κύκλο θα δοθούν οι λύσεις και επειδή αναφορά αναφέρεται σε αυτό το προσχέδιο του 2012 και εδώ έχει δρομολογηθεί ήδη ο δεύτερος κύκλος του σχεδιασμού, το είπε και η Κομισιόν, νομίζω ότι αυτή η αναφορά που έχει πλέον ε, καταστεί παροχημένη πρέπει να κλείσει. Και σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις, 25 υδρογραφικές λεκάνες έχει η Ισπανία σας προεδοποιώ λοιπόν, γιατί είχαμε ξαναπάει στον Εύρο το 2006 νομίζω εγώ ναι, ευχαριστώ να ξαναπάω. Αυτά που είπε συνέλεφος είναι πάρα πολύ ενισχυτικά. Τα είδα αυτό το 2006 και δεν έχουν λάβει και πολλά. Τι είναι παρηγοριά, πιο πολύ τώρα πια πριτανεύει η ανησυχία το τι θα γίνει. Μα, μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι δεν είναι σαφές, τι γίνεται με τα μέτρα, τι, γίνεται με το, επίπεδο του νερού, τι γίνεται με αυτές τις ε, τεχνητές λεκάνες υποδοχής των υδάτων, τι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε και αφού δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Μα είναι τρομερά, πολύ τρομερά αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δικαιολογεί αυτό που μας είπε προηγουμένως για τα υδρολογικά έργα στην Ισπανία και έχω τώρα κατά νου και τον Εύρο, αλλά το, πρόγραμμα, το πρόβλημα τελικά είναι συστημικό και διαρθρωτικό και συστηματικό δηλαδή ότι συνέχεια το πρόβλημα επιστρέφει, επαναλαμβάνεται. Οπότε έχουμε αυτή την αρνητική εμπειρία τόσων ετών, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία, πίστη, ελπίδα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο για να ανοίξουμε καινούργιο. Θα ήταν γελίο. Και αυτό σας λέω, νομίζω ότι όχι μόνο πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά, αλλά να ζητήσουμε την αποκατάσταση του Ισπανικού κράτους για όλα αυτά τα οποία ε, έχει πράξει και είναι αντίθετα με κάθε νομοθεσία. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται ο κατάλογος των προσώπων που είχα σημειώσει. Είμαι βέβαια ότι αν προχωρήσω μέσω να δώσω το λόγο στην αναφερομένη, γιατί ακούσατε ορισμένου από τους βουλευτέ που έλαβαν το λόγο. Ε, αν θέλετε να ξαναλάβετε το λόγο, κυρία Ματρίντε Φοντέν, έχετε το δικαίωμα αυτό. Ναι, θέλω να απαντήσω στον κυρία Γιούσο. Πράγματι, μιλάμε για το δρολογικό σχέδιο που εγκρίθηκε το 2014. Αυτό συζητούμε τώρα, αυτό είναι στο τραπέζι. Είπαμε όμως επίσης ότι βασιζόμαστε και στην αναθεώρηση αυτού του δρολογικού σχεδίου που είναι ουσιαστικά ακριβώ το ίδιο με το προηγούμενο, που εγκρίθηκε πέρυσι δηλαδή. Από αυτή την αφετηρία κινούμε λοιπόν και 30 ε, Ιουνίου λίγη περίοδο περίοδος που μπορούμε να καταθέσουμε τις καταγγελίες και θα το κάνουμε εμείς, είναι σαφές ότι αν αυτό το αναθεωρημένο σχέδιο είναι το ίδιο με αυτό το υδραυλικό σχέδιο που εγκρίθηκε πέρυσι, δεν έγιναν και πολλές τροποποιήσεις. Αυτό που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε είναι τι θα γίνει μέχρι τα τέλη του έτους, οπότε και θα εγκριθεί αυτό το υδραυλικό σχέδιο. Αυτό που έχουμε όμως στο τραπέζι αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχαμε πέρυσι. Συνεχίζουμε λοιπόν να μην ξέρουμε πώς έχουν τα υδάτα, τι κατάσταση έχει μάθει των υδάτων. Έχουμε τα 405.000 εκτάρια των αρδευόμενων εκτάσεων. Έχουμε ακόμη... Για να τα βρω. Τέλος πάντων, μην τα ξαναλέω, τα είπα. Τίποτα δεν άλλαξε. Στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε. Και γι' αυτό ε, εμείς ε, αυτό καταγγέλουμε. Ότι το σχέδιο του Ρολικού είναι το ίδιο με αυτό που εγκρίθηκε πέρυσι. Thank you very much. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Προτείνω τώρα το εξή επί της ε, συγκεκριμένη αναφοράς. Να διατηρηθεί ανοιχτή. Αυτό άκουσα άλλωστε από τους συναδέλφους. Και επιθυμώ να στραφώ τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στις ε, Ισπανικές αρχές, τους προσώπους των Ισπανικών αρχών που είναι παρόντες. Παρακαλώ να προετοιμαστείτε για να συναντηθείτε ξανά μαζί μας και να μας υποβάλλετε πληροφορικά στοιχεία για ενημέρωση πριν να προχωρήσουμε στην επιτόπου αποστολή των αρχών του επόμενου έτους. Να είστε έτοιμες ή έτοιμοι να προσέλθετε εφόσον σας προσκαλέσουμε και να παράσχετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που θα διαθέτετε στην γραμματεία της Επιτροπής μας. Αυτά μπορούμε να κάνουμε για την ώρα. Κατανοώ καλά από την συγγύη σας αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ότι συμφωνούμε. Μάλιστα. Το επόμενο θέμα που έχω είναι το υπαριθμόν 7 για δραστηριότητες οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αποξήρανση της κήτης του ποταμού Χαράμα κοντά στη Μαδρίτη και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι προστατευόμενες περιοχές εκεί. Είναι μια παλιά αναφορά που έχει τον αριθμό 0804 του 2006. Ο Μιγγέλ Άνχελ Σάντσες Πέρες είναι παρόν και είναι αναφερόμενο. Έχετε το λόγο κύριε. Muchas gracias, eh, Presidenta. Eh, leo esta petición. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σα διαβάσω ε, την αναφορά αυτή από πλευρά των ε, συναγωνιστών μου. Αυτή η διαδρομή ξεκίνησε το 2006, φαίνεται παλιά υπόθεση. Όμω, αυτή η κατάσταση που διαπιστώνεται είναι η ίδια που ισχύει σε οποιοδήποτε ποτάμι. Σε αυτή μιλάμε για τη λεκάνη του τάγου. Είχαμε το σχέδιο του 2014 που ε, δεν εφαρμόστηκε, δεν είχαμε καμία αλλαγή από το 2006. Μία σας διαβάσω αυτό το κειμενάκι που μου έχουν δώσει οι συναγωνιστές μου. Ακριβώς όπως είπαν και οι συναγωνιστές για τον Γουαδιάνα ή για τον Εύρο, για τον Καστρίλ. Γιατί αυτά γίνονται ακόμα και στις Βαλιαρίδες και σε άλλα ποτάμια. Θα προτιμούσαμε να μπορούμε να απολαύσουμε το περιβάλλον, τα ποτάμια μας και να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες απειλές και όλα αυτά τα έντονα προβλήματα. Για να σας πω ποιο είναι το κείμενο που συντάξαμε. Αύγουστο και 2006. Για πολλά χιλιόμετρα έμεινε ξερός ο ποταμός Χαράμα. Κάπου στη μέση τη δρομή του. Είναι κοντά στην Μαδρίτη και αυτό έγινε γιατί δεν υπήρχε σωστή διαχείριση της ε, λεκάνης αυτής. Ήταν υπεύθυνη μια, ένας φορέας τέλος πάντων ε, δημοτικός. Και αυτό έγινε γιατί δεν υπήρχαν οικολογικές ροές από τον Βάδο και τον Αταθάρ που είναι παραπόταμος του Λοθόγια και, και όλα αυτά τα είδατα θεωρητικά πέφτουν στον χαράμα. Οπότε είχαμε μόνο 104 λίτρα ανά δευτερόλεπτο ως ροή από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Και αυτά τα, νερά, αυτές οι ροές ήταν ανεπαρκείς για να μείνει σε κάποιο ανοιχτό επίπεδο το νερό στο ποτάμι. Οπότε δεν υπήρχε το ελάχιστο απαραίτητο. Και πέσαμε τα 0 λίτρα ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή τίποτα. Και αυτή η αποξήρανση έφυξε όλη αυτή την ε, λεκάνη των ποταμών Χαράμα και Ενάρες. Η διοικητική αρχή της περιοχής της Μαδρίτης έδωσε προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα και στη σωτηρία των οικοσυστημάτων της περιοχής. και οργανώθηκε επομένω ένα δίκτυο για αυτού τους δύο ποταμούς. Πρόκειται για ένα χώρο 65 χιλιόμετρων και αυτό το δίκτυο απορροής ήταν όλα αυτά τα χιλιόμετρα και πρόκειτο και για κάποιους παραποτάμους που είχαν χαρακτήρα όμως εποχιακό. Ε, το φυσικό περιβάλλον εκεί είχε θεωρηθεί ότι είναι προτεραιότητα να προστατευτεί. Είπαμε επίσης ότι υπάρχουν και άλλες προστατευόμενες περιοχές κοντά στο ποτάμι καταγεγραμμένες περιοχές και Τα ζητήματα είναι τα εξή. Ότι είχαμε τώρα σιγά σιγά μια επιδείνωση αυτού του περιβάλλοντος. Και το 2006 έγινε κάποια προσπάθεια ρύθμισης. Οπότε υπήρχε μεγάλη πίεση επί του περιβάλλοντος λόγω αυτών των έργων. Και όπως είπαμε προηγουμένως, στον ποταμό Χαράμα είχαμε πάρα πολλά ε, είδη τα οποία πρέπει να προστατευτούν και τελευταία οι αρμόδιες αρχές προσπάθησαν να προγραμματίσουν το πώς θα γίνει διαχείριση των υδάτων και του περιβάλλοντος εκεί. Τώρα δεν έχουμε ένα αποκρισταλωμένο καθεστώς όσον αφορά το ροή των υδάτων στον λοθόγειο στον Χαράμα παρά το, τα σχέδια διαχείρισης. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα τηρηθεί αυτό το καθεστώς το οποίο προβλέπει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όπως επίσης και της πανίδας. Έχουμε εκεί μια σειρά φραγμάτων επίσης, τα οποία εμπλέκονται στο πρόβλημα. Υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τον όγκο των ροών του ύδατος, αλλά επίσης το πρόβλημα είναι και ποιοτικό. Και τι γίνεται, όταν διακόπτεται η ροή σε ένα ποτάμι, τότε είναι μεγάλη η ζημιά που προκαλείται ακριβώ όπω έγινε το 2006 στον ποταμό Χαράμα. Ευχαριστώ. Στρέφομαι πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οποίας εκπρόσωπος ε, κ. Ρομέρο εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ και να διατηρεί πνεύμα συνεργασίας. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο παράδειγμα αυτό, άλλη περίπτωση για το πόσο σημαντικό είναι να καταρτιστούν υδρολογικές ζωές οικολογικές ε, για να επιτευχθεί ο στόχος της καλής κατάστασης και η συντήρηση, η διατήρηση των προστατευόμενων ειδών και οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από το νερό. Το είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στην Ισπανία και πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρήσει ε, τις σχετικές διατάξεις για να τις προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητες των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από το νερό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επαρκή στοιχεία για να αφισβητήσει τα συγκεκριμένα, τις συγκεκριμένες ευρωλικές ε, ροές, αλλά μπορεί να αμφισβητήσει το ότι δεν είναι σχεδιασμένες οι μέθοδοι για να εγγυηθούν την ε, επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, όπως και των στόχων για τις προστατευόμενες περιοχές. Εξού και θεωρούμε ότι είναι δομικό το ζήτημα και άρα πρέπει να επιληθεί σε επίπεδο συνόλου των λεκανών απορροής. Thank you very much. Believe it or not, with 10 Spanish members. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, δέκα Ισπανοί συνάδελφοι που βρίσκονται εδώ δεν έχουν ζητήσει το λόγο. Α, βλέπω την κυρία Γιούσο τώρα, ζητεί το λόγο. Πρώτα όμως η κυρία Βαγίνα και μετά η κυρία Γιούσο. Τώρα άνοιξε το μικρόφωνο η ομιλήτρια. Θα ζητούσα ή θα πρότεινα τέλο πάντων ότι ενδιαφέρον θα ήταν η Επιτροπή μας να ζητήσει από το Δήμο της Μαδρίτης να εκπονήσει μια έκθεση, να ερευνήσει το ζήτημα. Δηλαδή, ποιες είναι οι υποτιθέμενες παράνομες ενέργειες οι οποίες έγιναν στο Δήμο της Μαδρίτης με το κανάλι της ε, Ισαμπέλης Δεύτερης. Καλό θα ήταν για να μάθουμε και λίγο περισσότερα πράγματα. Thank you, Mr. Κυρία εσείς. Και εγώ θα είμαι σύντομη, λέει η κυρία Αγίουσο. Μα λέει εδώ ετών ότι η εκμετάλλευση των υδάτων μέσω του διάβλου Ισαβέλ Β δεν προσφέρει τις απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπήρξε το σχέδιο το 6, το 14 αναθεωρήθηκε και λένε οι αναφέροντες ότι δεν υπάρχει τήρηση αυτών που προβλέπονται. Ναι, αλλά ε, δεν, είναι, δεν, είναι δεν, δεν είναι δυνατόν να μην τηρούνται αυτές οι διατάξεις γιατί έχουμε πολλή ξερασία και όλα αυτά εξαρτώνται από τις δημοτικές αρχές, είναι περίπλοκη η διαχείριση και η διοίκηση οπότε είναι δυνατόν να μην τηρούνται αυτά τα όρια οικολογικών ροών. Υπάρχει αναθεώρηση από την Επιτροπή των όσων προβλέπονται. Αλλά το θέμα είναι, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή κατά πόσον υπάρχει τήρηση αυτών των διατάξεων των οικολογικών ροών σε σχέση και με τον καιρό που επικράτησε το φθινόπωρο. Μα γίνεται να τηρηθεί όμως ό,τι προβλέπεται ε, γιατί ας πούμε στον Εύρο και όχι αλλού είχαμε σημαντικές πλημμύρες. That concludes uh, the... Εδώ εξαντλήθηκαν οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό μου, άλλος κανείς δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να πράξουμε είναι το εξής. Πρόκειται για μια παλαιά αναφορά που χρονολογείται το 2006. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δήλωσε, αν κατανόησα καλά, ότι έχει γίνει παραβίαση της κοινωνικής νομοθεσίας και δεν μένουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να έρθουμε σε επαφή με τον Δήμο Μαδρίτης για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση και να διαπιστώσουμε στην βάση των πληροφοριών που θα παράσχουν τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Έχετε άλλες προτάσεις εσείς, ε, συνάδελφοι. Δεν έχετε τίποτε άλλο να πείτε. Άρα δέχεστε την πρότασή μου. Αυτό να πράξουμε. Α, μπορούμε λοιπόν αυτό να κάνουμε τότε. Και Κύριε Μάτο. Μια ερώτηση. Δεν έχω πρόβλημα αυτό που προτείνετε, όμως δεν νομίζω ότι μπορούμε να απομακρυνθούμε από το πεδίο αρμοδιοτήτων μας. Ζητήθηκε εδώ να ζητήσουμε από ένα Δήμο να μας πει τι έγινε με το κανάλι της Ζαμπέλ, της Δεύσης κτλ. κτλ. Μήπως ξεπερνάμε τις αρμοδιότητές μας, δεν ξέρω. Η αρμόδια αρχή, ο Δήμος, ε, ε, δεν πρέπει να ερωτηθεί από την κυβέρνηση της Ισπανίας, όχι από εμάς, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι δικό, δική μας αρμοδιότητα να απευθυνθούμε απευθεία στο, στο Δήμο. Όχι ότι δεν λέω, όχι ότι λέω να μην ζητήσουμε πληροφορίες, απλά νομικά, ε, ποια νομική οδός, η νόμιμη οδός για μας. Peter ο κύριος Γιάρ. Ίσως η τον των συναδέλφων οφείλεται και σε μια μηχανία. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών διαπιστώσατε και η ίδια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δήλωσε ότι υπάρχει παραβίαση του κοινωτικού δικαίου, εξάλλου είναι και παλαιά η αναφορά. Έτσι λοιπόν η δική μου αυθόρμητη πρόταση θα ήταν ότι θα πρέπει οι αναφερόμενοι να έλθουν σε επαφή με τις ε, τοπικές αρχές εάν, να δουν εάν κάτι δεν πάει καλά με την εφαρμογή. Κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι μπορούμε να κρίσουμε την αναφορά. Οι αναφερόμενοι απευθύνονται στις τοπικές αρχές και εάν, διότι δεν απαγορεύεται κάτι τέτοιο, εάν υπάρξουν νέα δεδομένα μπορούν να επαναλάβουν την αναφορά. Και εγώ ε, αμφιταλαντεύομαι λίγο. Από τη μια μεριά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχει παραβίαση τη κοινωτική νομοθεσία. Από την άλλη μεριά οι αναφερόμενοι ε, είναι δυσαρεστημένοι. Αυτό δείχνει ωστόσο να έγκυται σε μια έλλειψη επικοινωνία μεταξύ των αναφερομένων και των τοπικών αρχών. Κάτι που νομίζω εννοεί και ο κύριο Μάτο. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί εδώ από τι Βρυξέλλες. Είναι κάπω περιορισμένε οι ε, μα. μας. ότι έχει δίκιο ο κύριο Μάτο. Ε, για να δούμε τώρα από αυτά που είπαμε πώς μπορεί να φτιάξει κάποιο συμβασμό η Πρόεδρος. Η Πρόεδρος. Έχετε δίκιο. Δεν έχει την αρμοδιότητα ωστόσο ο Δήμος Μαδρίτης για να ειδεί εάν έχει παραβιαστεί κάποια κοινωτική νομοθεσία ή όχι. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάλογο με τις Ισπανικές Αρχές. Δηλαδή την κυβέρνηση και τις άλλες ενδεχόμενες αρχές που εμπλέκονται. Τώρα, εγώ Αντιλαμβάνομαι ότι δεν σα έδωσα ξανά το λόγο, κύριε Αναφερόμενη. Έχετε λοιπόν το λόγο. Α, σας ευχαριστώ. Ήθελα απλά να διευκρινίσω κάτι που είπατε. Οι αρμοδιότητε για τη διαχείριση είναι κρατικέ στην Ισπανία. Το κράτο λοιπόν είναι το αρμόδιο. Η Ισπανική κυβέρνηση λοιπόν εφαρμόζοντας την οδηγία πλαίσιο, πρέπει να υποχρεώσει ή τέλος πάντων να δημιουργήσει ένα καθιστός ε, ροών, ροικών κατάλληλων, για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι, αν καταλαβαίνω καλά κύριε Μάτο, λέτε ότι πρέπει να τα αφήσουμε εντός τα προβλήματα, να τα μαζέψουμε και να τα εξετάσουμε στη χώρα μας. Αν όμως ε, κάνει ό,τι θέλει μια επιχείρηση με ένα κομμάτι ε, της ε, ροής του τάγου, δεν είναι ένα λεπτό θέμα. Αν πρέπει να υπάρξει ένα καθεστώς υδρολογικών ροών με βάση υδρολογικά υδρομορφολογικά δεδομένα, τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να δει κατά πόσο έχει γίνει σωστά η δουλειά και αν αυτές οι ροές είναι κατάλληλες για να προστατεύουν τα, τους υδροβιοτόπους. Και είπε και η κυρία ότι η Ισπανία έχει περίοδους ξηρασίας, ε, μεγάλης διάρκειας και επειδή είναι και η θερινή περίοδος, οι ζέστες κρατάνε μήνες, ε, πρέπει να δούμε σε ό,τι αφορά τις οικολογικές ροές έγιναν σωστά τα πράγματα με τις μεθόδους που χρησιμοποίησε η Ισπανία. Βγαίνουν τα νούμερα, είναι τα σωστά. Αυτό θα αποφασιστεί τώρα. Εδώ λέμε όμω ότι αποξηρέονται ποτάμια, μεγάλα ποτάμια, που γύρω του υπάρχουν προστατευόμενες από οδηγίε. περιοχή. Άρα κάποια αρμοδιότητα έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την προκειμένη περίπτωση για τον ποταμό Χαράμα. Η διαχείριση γίνεται από το κράτος, αλλά η διαχείριση του νερού της κοινότητα τη Μαδρίτης, του της Μαδρίτης, οφείλεται στο ότι Υπάρχουν, υπάρχει ένα μεγάλο σύστημα, ε, ένας ταμιευτήρας που είναι η λεκάνη του τάγου και μικρά συστήματα. Πρέπει να μπει μια τάξη. που θα βασίζεται στον κοινό νου και στο κοινό συμφέρον για να έχουμε όλοι νερό. Και να υπάρχει και, νερό βέβαια και για, τα οικολογικά, για τις οικολογικές υδρολογικές ροές. Okay. Η πρόεδρος, ωραία. Αρχίζουμε τώρα βέβαια ε, και καθυστερούμε λίγο χρονικά. Θα προτείνω λοιπόν το εξή. Να στείλουμε επιστολή στις Ισπανικές Αρχές και να τους ερωτήσουμε εάν όντως έχουν επιτευχθεί οι οικολογικοί στόχοι στο προκειμένο αυτό πλαίσιο. Αυτός θα είναι ένας τρόπος για να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση από τις ε, ορθές προβλεπόμενες αρχές. Δεν άκουσα βέβαια και κανέναν άλλο να κάνει καμιά άλλη πρόταση. Συμφωνείτε, λοιπόν. Ωραία λοιπόν. Θαυμάσια. Τότε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξή μα. Την 0748 του 2007 για υδρολογικά έργα στον ποταμό Καστρίλ στην Ανδαλουσία καθώς και άλλη αναφορά του 2007 για τις, τις ε, επιβλαβείς ε, επιπτώσεις έργων που προβλέπονται στον ποταμό Καστρίλ και ο αναφερόμενος Μιγγέλ Άγχελ Όρτης είναι παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβετε για ποιο μέρος σας μιλάω ποταμός Καστρίλ βέβαια είναι ένας μικρός ποταμός, έχει όμως μεγάλη οικολογική σημασία και μεγάλη σημασία ε, για τους γύρω πληθυσμούς. Και πριν ξεκινήσω θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί εργάζεστε για τα συμβάντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες πολλές φορές εμείς είμαστε απροστάτευτοι απέναντι στις κυβερνήσεις των, απέναντι των κυβερνήσεών μας που δεν α, θέλουν να υπερασπιστούν τελικά τα γενικά συμφέροντα πολλέ φορέ, αλλά παρασύρονται από τι ειρήνε ε, τη πρωτεύουσα και δεν του ενδιαφέρουν ε, αυτά που αποτελούν πραγματικέ μα ανάγκε και τα οποία ζητούμε κάθε μέρα, χωρί να σκεφτόμαστε το μέλλον. Γιατί κάθε μέρα, κάθε φορά που καταστρέφεται ένα ε, τοπίο, καταστρέφεται, ε, η ανακοσύστημα καταστρέφεται μέρος της ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν ξαναζητάμε την υποστήριξή σας για να αποφευθεί αυτή η αχρίαστη οικολογική καταστροφή που θα είχε μεταφορά τον από τον ποταμό Καστριλ. Δεν είναι η πρώτη φορά που απευθυνόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Αναφορών με μια καταγγελία για να παρασπιστούμε τον ποταμό Καστρίλ. Ίσως ε, έχουμε την αμφίβολη τιμή να έχουμε στη γη μας την αρχαιότερη ε, αντιπαράθεση όλων. Ήδη από το 16ο αιώνα ζητεί το εκτροπή από την ε, λεκάνη του ποταμού Καστρίλα στο βασίλειο τότε της Μούρθια. Και το 1774 και το 1816 και το 1926 έγιναν ε, διαδοχικές προσπάθειες εκτροπής αυτών των υδάτων. Τελευταία φορά που έγινε αυτή η διαπροσπάθεια να φύγουν, να φύγουν τα νερά από το εσωτερικό προς τις ακτές έγινε το 1986 ε, για να αναπτυχθούν ε, υποδομές, θερμοκήπια, γκολφ ε, και άλλες περιοχές αναψυχής. Έγιναν λοιπόν κάποια έργα για τη συλλογή του ύδατο από τις εκβολές του ποταμού, αλλά από την πηγή του ποταμού στο νερίο, στον ποταμό Γουαρδάλ, να φτάσει στι οριστέ του Καστρίλ. Καταθέσαμε τότε μία ε, καταγγελία, ε, τα κοινωνικά κινήματα. δικαιώθηκαν τα κινήματα και τα αιτήματά μας. Ε, το 2002 έγινε μια νέα προσπάθεια εκτροπής για να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση το νερό. Κατα... Φύγαμε πάλι στην Επιτροπή σας, την Επιτροπή Αναφορών, με άλλη καταγγελία και συνεπή αυτής της, ε, αυτού του διαβήματος παρέλυσε αυτό το σχέδιο, σταμάτησε η Ισπανική κυβέρνηση. Το 2007 τώρα ερχόμαστε ε, με τη σημερινή μας αναφορά, τη σημερινή καταγγελία. Είχε προηγηθεί με ένα βασιλικό διάταγμα κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκατης ανάγκης λόγω ξηρασίας. Ο στόχος ήταν να μην τηρηθεί πρώτον το δικαίωμα για την ενημέρωση της κοινή γνώμη και συμμετοχή των πολιτών σε τέτοιου είδους έργα. Σήμερα είμαστε εδώ λοιπόν για να κατηγορήσουμε, ε, να καταγγείλουμε μάλλον το παράλογο αυτού του έργου, το ότι δεν χρειάζεται να γίνει και αντικρούμε και τις ε, εκθέσεις με τις οποίες προσπαθεί να αιτιολογήσει την εκτροπή αυτή η Ισπανική κυβέρνηση. Το μόνο το οποίο λέγεται σε αυτές τις εκθέσεις είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ότι θα γίνουν κάποια έργα και κάποια ε, μεταφορά εδάτων που όχι απλά δεν είναι ε, κάτι που πρέπει να γίνει, είναι και παράνομο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Και έχουμε δώσει πρόσφατα και κάποια στοιχεία Έχουμε τις νομικές γραμματεύσεις του δικηγόρου μας και έχουμε και μία μελέτη του Πανεπιστημίου της Γρανάδα που βεβαιώνει τις απόψεις μας. Από την πλατφόρμα της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, καταφέραμε στο το δικαστήριο να ακυρωθεί αυτοδικαίως αυτό το διάταγμα περί ξηρασίας, ε, διάταγμα για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκηρύχθηκε παράνομο. προσπαθεί τώρα η κυβέρνηση με μια άλλη διάταξη για στο πέστο του νόμου περιλημάτων να περάσει από τη Βουλή για να καλύψει ε, αυτά τα κενά. Να περάσει λοιπόν ένα νόμο για το οποίο έχουμε επίσης εμείς καταφύγει στο ανώτατο δικαστήριο. Μάλλον τέθηκε ζήτημα αντισταγματικότητας αυτού του νομοσχεδίου ε, και μέχρι να κηρυχθεί συνταγματικό ημί δεν σύστηκε το νομοσχέδιο αυτό. Εμείς είμαστε κατά λοιπόν των έργων για την έκτροπη του ποταμού Καστρίλ. Θέλουμε να αποσυρθεί οποιαδήποτε βοήθεια οικονομική δίνεται για την χρηματοδότηση των έργων αυτών και θέλουμε η Επιτροπή σας να από την Ισπανική κυβέρνηση να εφαρμόσει την τελευταία απόφαση του δικαστηρίου. Να επιστρέψει τη γη στους κατόχους της, να αποκαταστήσει την περιβαλλοντική ζημία και να τηρήσει ευρωπαϊκές οδηγίες για το περιβάλλον και για τα ύδατα. Και θέλουμε να σας δείσουμε να διατηρήσετε ανοιχτή την αναφορά μέχρι ό,τι αποφανθεί το συνταγματικό δικαστήριο και να σας πω ότι θα πρέπει να προσαρμόσει τα υδρολικά της σχέδια Ισπανία σύμφωνα με τις διατάξεις ε, της οδηγίας πλαισίου για τα Να σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες ε, του υδρολικής λεκάνης του ποταμού Καστρίλ. Ζητούμε να ληφθεί υπόψη ο ποταμός Καστρίλ και ολοκληρώνω ή μάλλον ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ πολύ. το συγγνώμη, αλλά κάπως λίγο τα έχασα, γιατί πραγματικά με συγκινεί πολύ αυτό το θέμα. Thank you very much. And you have Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ, σας καταλαβαίνω. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να σας δώσω και να σας δώσω το λόγο δηλαδή πολύ περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάντως που ήρθατε και μας παρουσιάσατε τις εμπειρίες σας. σχετικά με την κατάσταση του ποταμού, καθώς επίσης και το τι σημαίνει για τη ζωή των περίοικων. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εάν είστε κουρασμένος κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής, ένας από τους βοηθούς μας θα σας φέρει ένα καφέ. Αυτή η αναφορά επίσης σχετίζεται με το θέμα της οικολογικής στάθμης των οικολογικών ροών ακριβώς όπως ε, συζητήσαμε για τις προηγούμενες αναφορές. Σε αυτή την περίπτωση κάναμε κάποια αξιολόγηση της τεχνικής μελέτης όπως μας την διαβίβασε ο αναφέρον και καταλήξαμε στο ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους ε, αρνητική επίπτωση από το έργο στον ποταμό Καστρίλ. επίση υπόψη το έγγραφα από τις αρμόδιες πανικές αρχές και την ανάλυση που έκαναν αυτές οι αρχές. Έχουμε όλα τα στοιχεία επομένω με τα οποία νομίζω ότι μπορούμε να στηρίξουμε την άποψη των αρχών. Πάντως, Βεβαίως έχει, έχουν επιληφθεί τα εθνικά δικαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εφαρμόσει το κινητικό δίκαιο. Επομένως, εκκρεμωδική ακόμα η υπόθεση. Οπότε και εμείς αναμένουμε τη σχετική απόφαση. Thank you very much. This was exactly the information. Ευχαριστώ. Αυτές τις πληροφορίες πραγματικά ε, έψαχνα και σας ευχαριστώ που μας τις παραχωρήσατε. Και τώρα παρακαλώ οι συνάδελφοι για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση και πρώτη η κυρία Γιούσο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Για άλλη μια φορά όπως προείπα. Αυτές οι τρογραφικές λεκανές είναι 25 και είναι αρμοδιότητα των διοικητικών αυτών περιφερειών και άλλες 13 που είναι αρμοδιότητα των κεντρικών αρχών, των κρατικών. Ο Γουαδαλκιβίρ είναι πάντως αρμοδιότητα της αυτόνομης κοινότητας συναδελφίας και όπως είπε ο αναφέρον, θα πούμε λίγα λόγια, το 2005 είχαμε αυτό το βασιλικό διάταγμα για την ξερασία και δυνάμει αυτού του διατάγματος η κυβέρνηση αλλά και η, αυτόνομη κοινότητα που ανήκαν στο ίδιο κόμμα ξεκίνησε αυτό το έργο. Ήταν και οπότε στη συνέχεια τα δικαστήρια απεφάσισαν ότι ήταν ε, παράνομη ενέργεια. Επομένως υπήρξε εδώ δαπάνια και διασπάθηση των δημοσίων χρημάτων. Μια που τώρα. Ε, γιατί είπαμε επομένως ότι δεν έγιναν αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν, οπότε 2005 μέχρι το 2010 συνεχίστηκαν τα έργα αλλά είπαμε ότι τότε δεν υπήρχε πρόβλημα παροχής υδάτων προς τις κοινότητες που όφυλαν να ε, δεχθούν τα ύδατα από αυτό το έργο. Έχουμε ομένω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και προκειμένου έχει δίκιο φέρω ότι θα πρέπει να ε, σταματήσει το, το, το σχέδιο, το πρόγραμμα αυτό και να ληφθούν υπόψη τα όσα έχουν πει οι Ισπανικές αρχές, αυτές οι μελέτες που υπέβαλαν οι αρχές. Δεν ξέρω τι ημερομηνία φέρουν αυτές οι, αυτά τα υπομνήματα, αυτές οι μελέτες των Ισπανικών αργών. Η κυρία Βαλίνα. Έχει δίκιο ο αναφέρον. Αλλά και οι υπόλοιποι δεν είναι δυνατόν να κρυθεί μια ένσταση, μια καταγγελία ανάλογα με το ποιος, ποιο κόμμα έχει την ανάλογη κοινότητα ή την ε, κυβέρνηση. Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες, θα πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, θα προστατεύουμε τον, τον κόσμο και την ε, φυσική εθνική μας κληρονομιά άσχετα με το ποιος βρίσκεται στο πιδάλιο. Πρώτη επομένως για άλλη μια τέτοια περίπτωση. Εν προκειμένου και όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχουν στοιχεία. Διαπιστώνουμε πάντως μελετώντας όλες αυτές τις αναφορές ότι το πρόβλημα είναι συστημικού, δομικού, διαρθρωτικού χαρακτήρα οπότε δεν έχουμε τα στοιχεία. Να δούμε τι θα κάνουμε. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Να δούμε τι θα κρίνουν τα δικαστήρια μέχρι ότου όμω ληφθεί κάποια δικαστική απόφαση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέξει τι πληροφορίε που πρέπει. Επομένω, ανοιχτή αναφορά και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Κυρία Καμπεθόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να πω αυτό που είπε στην αρχή και η κυρία Δαλίνα. Εγώ είμαι υπέρ τη βιωσιμότητα και να εγγυηθούμε ότι η οι διατάξει την εφορία του περιβάλλοντο, όποιο και αν είναι στην εξουσία. Και για το συγκεκριμένο θέμα τη αρμοδιότητα για το Γουανταλκιβίρ, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση. Θα μπορούσα να σας αναφέρω την απόφαση την πρόσφατη του συνταγματικού δικαστηρίου γιατί καταγγέλθηκε το τελευταίο εγκεκριμένο καθεστώς της αυτονομίας. Για το που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Εγώ ε, να λαμβάνω αυτό που είπα από την αρχή, ότι υπάρχει πρόβλημα ουσίας εδώ. Και έχει δώσει κάποιες απαντήσεις κομισιόν το 11 και εκεί βλέπω ότι το πρόβλημα είναι και εδώ η έλλειψη υδρολογικών σχεδίων και η ανεπάρκεια αυτών των προγραμμάτων. Ε, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δεν ξέρω ποιο είναι υπεύθυνο, ποιο πρέπει να απαντήσει. Αυτό που συζητήσαμε από την πρώτη αναφορά το συζητάμε και τώρα. Λαμβάνοντα υπόψη ότι σε άλλε περιπτώσεις εδώ, όταν το θέμα που θεωρούσαμε ότι έχει κριθεί, ε, το έχει, ε, έχει πλέον δικαιοσύνη, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και καλό είναι να ζητήσουμε και από την κυβέρνηση της Ανδαλουσίας να μας δώσει ή να κάνει μια έκθεση για να δει που βρίσκεται η κατάσταση. Ή ε, τέλο πάντων η Ισπανική κυβέρνηση, αν όχι η αυτόνομη κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς συμβιλογνώμων για να κατανοήσει τις καταστροφές που θα προκληθούν από μεταφορά της κήτης του ποταμού. Υπάρχουν πολλές ωστόσο σκιές μέσα σε αυτό το ντοσιέ. Προφανώς η ισπανική δικαιοσύνη ακόμα δεν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της, οφείλουν να αναμένουν την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Εγώ προτιμώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και συνολικά θα ήθελα να πω, επειδή είδαμε έναν αριθμό αναφορών να υπάρχουν και άλλες, είναι πρόβλημα εθνικό. Είναι Βεβαίω γεγονό ότι έχει ένα πρόβλημα βρόχομετρία η Ισπανία όντω αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό η Ισπανία αλλά το γεγονό ότι υπάρχει πρόβλημα εξηρασίας δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστρέψουν το υπόλοιπο περιβάλλον. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Πώ μπορεί η Ευρώπη να ενισχύσει την χώρα αυτή, να ε, βοηθήσει με κάποιο τρόπο, δεν είναι βέβαια μονάχα οι ε, τοπικές αρχές που θίγονται, και οι τοπικές αρχές και οι μη κρατικέ οργανώσεις και όλοι όσοι ζουν χάρη στους ποταμούς αυτούς πρέπει να μπορέσουν να βοηθούν. Και εκεί έχει μια ευθύνη και η ίδια η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος και τώρα ο κύριος Ορτσίθ Λόπεθ. Δεν έχω πολύ χρόνο, ε, όπως είδατε και δεν μπορούσα να εξηγήσω ακριβώς τέσσερα. μας. Πρέπει να σας πω ότι για το Γουαλταρκιβίρι η αρμοδιότητα την έχει κεντρική κυβέρνηση. Και θέλω να πω επίσης ότι εμείς θα θέλαμε σε αυτή την περίπτωση να επεκτείνουμε αυτή την καταγγελία για τετραλογικά σχέδια τα οποία καταρτίζονται και στον πρώτο κύκλο και στο δεύτερο. Εμείς συμμετείχαμε στη διαδικασία και κάναμε κάποιες καταγγελίες και διατυπώσαμε τις ε, ενστάσεις μας και ότι παραβιάζεται δηλαδή η Ευρωπαϊκή Οδηγία και ότι δεν μας προσέχουν. Έχουμε καταθέσει μελέτες από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας ε, και άλλες ε, και άλλα στοιχεία που δείχνουν πόσο ευαίσθητος είναι ο ποταμός και η οικολογική ροή που θα αφήσουν θα είναι πάρα πολύ αβαθής. Εμείς είμαστε και στην φάση που εξετάζουμε το δεύτερο δολογικό σχέδιο που θα έχει κατατεθεί μέχρι τα τέλη του Ιουνίου και φοβούμε πολύ ότι δεν θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Θα σας ε, παρακαλούσα λοιπόν να αποφεληθείτε τις επίσκεψή σας στην Ισπανία, να επισκεφτείτε και άλλες περιοχές για να καταλάβετε πολύ καλά το πρόβλημα το οποίο σας ε, αναφέρουμε εδώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Πολύ ευγενική. Σας βεβαιώνω ωστόσο ότι αρχάς του επομένου έτους όταν θα κάνουμε την αποστολή δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να φτάσουμε μέχρι τη Γρανάδα διότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ περίπλοκο αλλά ίσως βεβαίως κοιτάξτε μεμονωμένα οι βουλευτές μπορούν να ταξιδέψουν μπορείτε ενδεχομένως να προσκαλέσετε ορισμένους από τους Ισπανούς Ευρωβουλευτές να προσέλθουν να δουν οι ίδιοι ή και βουλευτές από άλλες ε, χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ε, δυνατότητα που έχουν να ταξιδέψουν και να πάνε να δουν οι ίδιοι περί πρόκειται. Σας βεβαιώνω πάντως ότι η Επιτροπή Αναφορών θα συνεχίσει να εξετάζει το θέμα. Και επειδή τώρα είναι βέβαια η υπόθεση ενώπιον Εθνικού Δικαστηρίου στην Ισπανία, εγώ θα προτείνω να μείνει η αναφορά ανοιχτή μέχρι ότου εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό που θέλω επίσης να προτείνω είναι να γράψουμε ε, να γράψουμε στις ανδαλουσιανικές αρχές να θέσουμε υπόψη τους, δηλαδή να τους υπενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή Αναφορών ε, παρακολουθεί το θέμα. Ίσως είναι χρήσιμο αυτό. Και οι Ισπανικές αρχές που είναι παρούσες σήμερα να αντιληφθούν ότι είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και σοβαρά. Και βεβαίως θα επανέλθουμε όταν θα εκδοθεί η απόφαση του Ισπανικού Δικαστηρίου. Και βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλαξη των συνθήκων παρακολουθεί το θέμα και θα μας ενημερώσει ξανά, ξανά όταν θα απαιτείται. Ε, συμφωνείτε, νομίζω λοιπόν ότι συμφωνείτε και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διατάξεως. Έχουμε κάπως αργοπορήσει ήδη η επόμενη έκθεση επίσης ισπανική βεβαίως του Συνδέσμου Διαχείρισης υδρολογικού Σχεδιασμού του Άρτο Γκουαντιάνα και είναι υπαριθμόν 1957 του 2012. Ο αναφερόμενος ή οι αναφερόμενοι δεν είναι παρόντες, εκπροσωπούνται όμως από τον Μαριάνο Βελάσκο Λισάνο. Μάλλον σημαίνει την κυρία ε, Βελάσκο Ρισιάνα. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Pues, eh, buenas tardes, muchísimas Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε που μας ε, ακούσατε. Εκπροσωπώ τον αναφέροντα για τον Τάγο. Αλλά επίσης θα μιλήσω τώρα και για τον Γουαδιάνα. Έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την διαχείριση των υδάτων, όπως ξέρετε, όπως συζητήσαμε ε, όλο το απόγευμα σήμερα και υπάρχουν κάποια γενικού χαρακτήρα ζητήματα για αυτές τις ε, λεκάνες υπόδειξη των υδάτων και επίσης έχουμε και θέματα ότι η περιμετάλλευση οδήγησε σε μόλυνση. Και ρίπανση λοιπόν στο μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα σχέδια για τις λεκάνες δεν οδηγούν σε κάποια λύση των σχετικών προβλημάτων. Επομένως, εάν εμείς δεν δούμε το πώς η οδηγία για τα ύδατα πώς θα υποστεί κάποια τροποποίηση για την αλλαγή της διαχείρισης εάν επομένως δεν κάνουμε σχετικές ενέργειες τότε μπορεί να έχουμε πάρα πολλά σχέδια για τις τεχνητές λεκάνες απορροής αλλά η κατάσταση θα μείνει αμετάβλητη. Ο Γουαδιάνα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Δεν περνάει από βουνά. Πρόκειται για ένα είδος ποταμού μοναδικού στην Ευρώπη. δεν πηγάζει από βουνό, αλλά από τον εντροφόρο ορίζοντα. Είναι αυτό που ονομάζουν ποτάμι που υπάρχει, σαν και αυτά τέλος πάντων, που υπάρχουν στην Λαμάντσα. Βεβαίω και υπάγεται στο δίκτυο Natura. Ε, προστατεύεται από τη σύμβαση Ράμσαρ και από άλλες ε, συμβάσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο το περιβάλλον εκεί και όπως είπαν πριν ε, πηγάζει, σχετίζεται ε, με τον υδροφόρο ορίζοντα. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Η υπερεκμετάλλευση. Κοιτάξτε αυτές τις φωτογραφίες. Η κάτω φωτογραφία προέρχεται τη δεκαετία του 50. Από αμερικανικές πηγές προέρχεται η φωτογραφία και η άνω φωτογραφία είναι περσινή. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, έχουμε αυτού του είδους τα ε, επίπεδα και τα οποία εξαφανίζονται από την ξηρασία μέσα σε μία τριακονταετία. Μιλάμε για 30.000 εκτάρια που έχουν ε, ε, καλυφθεί, που έχουν τελικά εξαφανιστεί μέσω της ε, ξηρασίας. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα και δεν μπορεί να λυθεί με τα υδρολογικά σχέδια. Βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα, στην πρώτη ε, στήλη, βλέπετε τα διαθέσιμα ύδατα. Αυτά τα οποία προέρχονται από την εντοφόρεζοντα κάθε χρόνο. Τώρα, όσον αφορά ε, τα δικαιώματα τα οποία εκχωρούνται ε, προς πότισμα, είναι στην δεύτερη στήλη. Δηλαδή πολλές φορές εκχωρούνται τα διπλάσια ή τα τριπλάσια. Και σε κάποιες περιοχές έχουμε πενταπλάσια άντληση, τέλο πάντων χρησιμοποίηση υδάτων για, ε, για από όσο νερό ρίχνει στο ποτάμι ο δροφός φορέσιντας. Επομένω δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά το ποτάμι. Γι' αυτό βλέπετε τι γίνεται με την πρώτη στήλη. Να, τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι ακόμα πιο ε, μικρά. Μετά έχουμε το τι προβλέπεται από το σχέδιο. Πρόκειται για κάποιον, κύκλο, για κάποια φάση που υπάρχει, δεν, δεν υπάρχει το υγρασία, αλλά είναι 37 παραπάνω. Επομένως αλλάζουν αυτά τα στοιχεία στο πρώτο σχέδιο και έχουμε αυτές τις ε, τιμές. Στο πρώτο, στην πρώτη εφάνεια, και εδώ στη δεύτερη έχουμε ε, αυτήν ε, τον υπολογισμό που είναι σκανδαλώδης. Ό,τι δηλαδή δίνεται για πότισμα ε, είναι πολύ περισσότερο από τα ύδατα, από τις δυνατότητες του υδροφόρου ορίζοντα. Γι' αυτό και φτάσαμε στην κατάσταση που αποτυπώνει στην πρώτη φωτογραφία. Πρόκειται για έναν ποτάμι ε, το οποίο το 2009 ε, ήταν έτσι από τη φωτογραφία. Αυτός είναι ο ποταμός Γουαδιάνα. Ενέτη 2009. Και βλέπετε αυτή την πινακίδα που λέει μην ε, βουτάτε, μην κολυμπάτε και βρίσκεται εν μέσω μιας περιοχής Κατάξερες. Για το 2009 εξαφανίστηκε το ποτάμι. Βλέπετε εδώ κάποια τυχώματα τα οποία συγκρατούσαν το ποτάμι, α, τώρα όμως είναι κατάξερο. Ο αριθμός των μετρητών, των των πηγαδιών που υπάρχουν στην περιοχή, είναι αβέβαιο γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικός ολοκληρωμένος έλεγχος λένε για 60.000 πηγαδία. Όμως δεν υπάρχουν ε, παντού μετρητές, οπότε είναι άγνωστο περί τίνος ε, ποσότητος μιλούμε. Άρα, το μεγάλο πρόβλημα είναι η υπερεκμετάλλευση, αλλά το δεύτερο είναι η μόλυνση. λόγω της γεωργίας υπάρχει παντού κάποια διάχυτη μόλυνση στον Ουαδιάνο. Με κόκκινο είναι οι πιο μορισμένες ζώνες. Είναι ακριβώς εκεί που έχουμε γεωργίες εκμεταλλεύσεις. Βλέπετε εδώ τις περιοχές που υπάρχει ο κίνδυνος της μεγαλύτερης ε, μόλυνσης. Και έχουμε επίσης αλλού έχουμε τη διάχυση της μόλυνσης και αλλού έχουμε σε συγκεκριμένα σημεία ε, τις μολυσμένες περιοχές. Η Πρόεδρος. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Τρίγκες Ρομέρο, έχετε το λόγο εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Εν προκειμένου η αρχική αναφορά αφορούσε την διάλυση του φορέα διαχείρισης του Άνω Γουαδιάνα. Οπότε έχουμε την ανακοίνωσή μας του 2014 που αναφέρεται ότι και εμείς θεωρούμε ότι εδώ τη συντρέχει περίπτωση παραβίαση της κοινωνικής νομοθεσίας. Τα δε μέλη είναι στη διακριτική του ευχέρεια το να λάβουν τα μέτρα, τα αναγκαία, ούτως ώστε να πετύχουν τους στόχους που έχει θέσει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, συμφωνούμε με τον προβληματισμό για την υπερεκμετάλλευση ε, του Άνω Γουαδιάνα. Και ακριβώς εδώ πέρα έχουμε διαχείριση πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με την υπόλοιπη Ισπανία και ισχύουν αυτό που είμαι και για τις άλλες ε, αναφορές. Όλα τα στοιχεία μας υπέβαλε ο αναφέρον. Τα έχουμε λάβει υπόψη. Και όλα αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν σε αυτή την οριζόντια ανάλυση που κάναμε για την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου. Έχουμε προβεί σε ανταλλαγή πληροφοριών με τις πανικές αρχές για το τι γίνεται στο ποτάμι αυτό, για το ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και ενημερωθήκαμε ενδελεχώς όσον αφορά την εκμετάλλευση και υπερεκμετάλλευση, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των υδάτινων πόρων. Ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο αναφέρον. Επίσης για το θέμα των μετρητών, για τον έλεγχο των υπογείων υδάτων. Και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα Όλα αυτά αποτελούν ζητήματα τα οποία παρακολουθούμε με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων. Επίσης, ζητήσαμε από τις Ισπανικές Αρχές να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους, τόσο ώστε να δούμε ακριβώς ε, ποια είναι η μετάλλευση των υδάτων και σε σχέση με το τι, ε, νερό επιτρέπουν να εκχωρηθεί, ούτως ώστε να υπάρχει αντιστοιχεία με τις πραγματικές δυνατότητες. Ακριβώ γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές απολύουν πάρα πολύ από τις πραγματικές δυνατότητες. Thank you very much and thank... Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστώ που υπήρξατε και τόσο σύντομος και ακριβής στην απάντησή σας. Τώρα, η κυρία Ιούσο. Ευχαριστώ πολύ. Για μια ακόμη φορά κυρία Πρόεδρε, φοβούμε ότι θα πρέπει να μεταφέρετε την έδρα της Επιτροπής σας ε, στην ε, Ισπανία λόγω του αριθμού των αναφορών που προέρχονται από τη χώρα μου. Η αναφέρουσα μας παρουσίασε μια αρκετά καταστροφική, θα τη χαρακτήριζα, κατάσταση. Πράγματι υπάρχει αυτή η επεκμετάλλευση, λόγω άρδευση, το γνωρίζω το μέρος, αλλά πριν από 20 χρόνια περίπου κυβέρνηση, για να μην λέτε ότι μιλάω για τις ε, κυβερνήσεις ε, που δεν είναι της δικής μου πολιτικής οικογένεια. Άρχισε λοιπόν να παίρνει κάποια μέτρα η τότε κυβέρνηση για αυτά τα φρεάτια και απέσυρε κάποιες ε, αρδευόμενες τάσεις. Στην Καστίγια Λαμάτσα τότε συζητούσαμε το θέμα των μετρητών μεταξύ άλλων. Καμία σχέση δεν έχει ε, το τι γινόταν ε, πριν 20 χρόνια και τι γινόταν πέρυσι. Πέρυσι είχαμε κανονικές βροχοπτώσεις και οι πίνακες είναι πάρα πολύ ωραίοι και η περιοχή είναι πάρα πολύ όμορφη ούτως ή άλλως. Το η πολιτικής σταμάτησαν να καλλιεργούν αραβόστο επειδή δαπανά πολύ νερό, ε, κατάλληλα πολύ νερό αυτή η μεταρρυθμιση της κοινης γεωρικης πολιτικης Σταμάτησα να καλλιεργουν αραβωστε επειδη δαπανα πολυ νερο καταλληλα πολυ νερο αυτη η καλλιεργεια Βέβαια δεν έχει καμία σχέση αναφορά με αυτό. Θεωρούν ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί το ρολικό σχέδιο επειδή αυτό το, αυτή η κοινοπραξία ε, διαλύθηκε. Αυτό όμως αποφασίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν ήταν ε, προαπαιτούμενο για το υδρολογικό σχέδιο. Και αυτή η κοινοπραξία ούτε καν έχει αρμοδιότητα για όλη τη λεκάνη απορροής, αλλά μόνο για το Άλτο Γουαδιάνα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ε, κοινοπραξία για να εφαρμοστεί αυτό το υδρολογικό σχέδιο. Επειδή λοιπόν αναφέρεται συγκεκριμένα ε, η αναφορά στην κοινοπρεξία, πιστεύω ότι πρέπει να κλείσει, γιατί έχει καμία σχέση η κατάσταση με τι αδερφόμε εκτάσεις και τι γίνεται με τον υδροφόρο ορίζοντα με, αυτό το, με αυτή την κοινοπραξία που διαλύθηκε ή δεν διαλύθηκε τέλο πάντων. Ευχαριστώ. Thank you very much. And on... Ε, σας ευχαριστώ πολύ. ποιος θα είχε αντίρρηση να μεταφερθεί η Επιτροπή Αναφορών στην Ισπανία βλέποντας εδώ τον γκρίζο ουρανό τι ωραία που θα ήταν να δούμε τη λιακάδα της Ισπανίας άλλος κανείς επιθυμεί να το λόγο κανείς θα δώσω τότε το λόγο πάλι στην αναφερόμενη σύντομα και αν μπορείτε να εξηγήσετε λίγο περισσότερο την επέκταση του πεδίο αναφοράς της αναφοράς σας ε, διότι αυτές οι πιο πρόσφατες πληροφορίες δεν, είναι, δεν ταυτίζονται με το αρχικό αντικείμενο της αναφοράς σας. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι όταν κατατέθηκε αυτή η αναφορά κατατέθηκε επειδή το ειδικό ε, υδρολικό σχέδιο για την Άλτα Γουαδιάνα και το συγκεκριμένο όργανο που θα διαχειριζόταν ήταν ένα εργαλείο για να αγοραστούν και να αφαιρεθούν αυτά τα δικαιώματα ουσιαστικά. Το θέμα της υπερεκμετάλλευσης είχε κάποια, υπήρχαν κάποια εργαλεία, μπορούμε να συμφωνήσουμε, είναι έγκυρα αυτά, και συγκεκριμένα ήταν η ανάθεση αυτή ε, σε αυτή την κοινωνία. Και πράγματι, κατατέθηκε αυτή η αναφορά διότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η ανάθεση με τον λόγο και της οικονομικής κατάστασης ε, στην Ισπανία τότε. Το πρόβλημα είναι όμως ότι εμείς δεν έχουμε πλέον αυτό το εργαλείο που είχαμε για να ρυθμίσουμε το ζήτημα. Εμείς θα θέλαμε να συνεχιστεί η αναφορά, να παραμείνει ανοιχτή, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε αυτό το εργαλείο που είχαμε στη θέση μας πριν. Και επειδή ε, σε αυτούς τους πίνακες βλέπετε την ε, συγκεκριμένη περιοχή είναι σε καλή φάση γιατί υπήρξε πραγματικά ένας ε, κύκλος ε, βροχοπτώσεων πολύ έντονος το 2009 μέχρι το 2012. Πάρα πολλές βροχοπτώσεις, αλλά φέτος δεν ήταν τόσο πολλές οι βροχές όπως το προηγούμενο έτος ή το προπροηγούμενο, άρα το πρόβλημα παραμένει. Διότι σε αυτό το πίνακα που σας έδειξα ισχύει το πρόβλημα. Παραμένει. Ευχαριστώ. Okay. Η Πρόεδρος. αντιλαμβάνομαι ότι το αρχικό αντικείμενο της αναφοράς δεν είναι πλέον τόσο ακριβές. Ακούσαμε την πρόταση να κλείσει η αναφορά. Μπορούμε να το πράξουμε αυτό και ταυτόχρονα να στείλουμε μια επιστολή στις αρμόδιες αρχές όπου τις ενημερώνουμε ότι ασχολούμεθα με αυτή την υπόθεση και βεβαίως πάντοτε μπορείτε να, θέσετε μια, να υποβάλλετε μια νέα αναφορά. Είστε σύμφωνοι. Ναι. Και Ματών εσείς. Η πρότασή σας έχει ενδιαφέρον. Αλλά εάν το κάνουμε αυτό, λύνουμε το πρόβλημα του τύπου, όχι όμως της ουσίας. Σύμφωνοι με την επιστολή, αλλά ίσως να δώσουμε περισσότερη έμφαση απέναντι στις Ισπανικές Αρχές στις ε, οικολογικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις τη υποθέσεω αυτή. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, πολύ σωστά. Ωραία, μπορούμε τότε να κάνουμε το εξή. Γράφουμε μια επιστολή όπου εξηγούμε και αναπτύσσουμε λίγο το θέμα και μετά κλείνουμε την. και τώρα μάλλον κλείνουμε την αναφορά. Εφόσον το πρόβλημα συνεχίσει να εμφίσταται, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να υποβάλλεται νέα αναφορά με ε, διευρυμένο αντικείμενο πλέον διευρυμένο από αυτό που ε, είχε η αρχική αναφορά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Το υπαριθμόν 10 τώρα. Είναι η 0459 του 2011 για τα νερά του ποταμού Τάχος που ε, πέφτει στον ποταμό Σεγούρα καθώς και με διάφορες ε, δομές σωλήνων. Ο αναφερόμενος δεν είναι παρόν, δίνω το λόγο ευθύς αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν είστε ε, ακόμα εδώ και δεν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα για να αναπαυθείτε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Πολύ σύντομα λοιπόν να αναφέρουμε την ανακοίνωση που είχαμε στείλει πέρυσι για την αναφορά αυτή. Από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτό το ε, σχέδιο, αυτό το έργο δεν εντάσσεται στο δρολικό σχέδιο του ποταμού Σεγούρα και εγκαταλείφθηκε. Άρα δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Uh, Η Πρόεδρος. Άρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έργο έχει διακυρωθεί. Και αυτό έχει κοινοποιηθεί και στον ίδιο τον αναφερόμενο με έτοιμα σχολείου εκ μέρους του. Δεν έχει ληφθεί καμία αντίδραση ως τώρα από μέρους του. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να κλείσει η αναφορά. Σύμφωνοι. Ωραία. Α, τώρα επιτέλου αρχίζουμε να κινούμεθα με μεγαλύτερη ταχύτητα δηλαδή ενώ προχωρούμε στο υπαριθμό 11 η 092114 κατά του υδρολογικού σχεδιασμού των Βαλεαρίδων νήσων. Βέβαια ο αναφερόμενος ή αναφερομένη είναι παρούσα, Μαρία Οχένια Πριέτο Ρουίς και... Α, πάλι εσείς. Μάλιστα, πάρετε το λόγο λοιπόν. Για άλλο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λυπάμαι, λυπάμαι που έχουμε γίνει βαρετοί ε, για το πρόβλημα των υδάτων στην Ισπανία, αλλά έχουμε σοβαρά προβλήματα σχετικά. Και μου είπαν οι συναγωνιστέ από τις Βαλίδε να σα εξηγήσω ότι γίνεται. ακριβώ όπως και στις υπόλοιπε τρολογικές λεκάνες έχουμε και εδώ υπερεκμετάλλευση αλλά και ε, μόλυνση. Και ούτε εδώ τα σχέδια αποτελεσματικά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Στις Βαλιαρίδες Υπάρχει πρόβλημα. Η υπερεκμετάλλευση που γίνεται ακόμα χειρότερη λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα του εδάφους. Παροξύνονται τα προβλήματα επειδή είναι νησιά. Αν βλέπετε από εδώ πέρα αυτό το χάρτη με τις ζώνες υπερεκμετάλλευσης. Και όταν έχουμε υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου ορίσαντα παραπάνω τις δυνατότητες, Έχουμε βάλει εκεί το κόκκινο χρώμα και, πορτο, και πορτοκαλί στις σχετικές ε, περιοχές. Εκεί, στο νότο, κυρίως της νήσου. Μιλάμε για 150% υπεράντληση. Και έχουμε κάποιες πολιτικές, δεν έχουμε πολιτική, συγγνώμη, μείωση των ε, δικαιωμάτων, ε, ούτε κανένα είδους ε, πρόγραμμα τοποθέτησης ε, μετρητών. Και αντλούνται όλο για περισσότερα ύδατα, περισσότερες γεωτρήσεις στη Μαγιόρκα. Η νομοθεσία επομένως δεν συγκρατεί τις νέες γεωτρήσεις. Άρα θα πρέπει να υπάρξει κάποιο τροπής νομοθεσίας για το πόσο κοντά είναι μία γεώτρηση το ένα πηγάδι τέλο πάντων από το άλλο. Να είναι από τα προβλήματα. Κατά μέσο όρο είναι 70 μέτρα βαθιά αυτά τα πηγάδια. Τώρα, το πιο σοβαρό πρόβλημα αφορά την κατάσταση των υδάτων. Η μόλυνση φτάνει σε κάποιες οριακές τιμές που οι οποίες είναι απαράδεκτες από τα 37 μιλιγκράμμ ανά λίτρο από αζωτούχα και φωσφορούχα έχουμε φτάσει τα 200 μιλιγκράμμ ανά λίτρο. Η τιμή των 37 είναι ο αποδεκτός μεσός. Επομένως έχουμε μεγάλη μόλυνση όλων των υδάτων. Αυτό από τα ζωτούχα λιπάσματα που αντιστοιχούν φυσικά στις γεωργικές περιοχές. Εκεί είναι η πιο μεγάλη μόλυνση. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Είναι το ότι από την εκμετάλλευση των υδάτων, ή μάλλον την υπερεκμετάλλευση, έχει μπει ε, θαλάσσιο νερό μέσα στον τροφέρο ορίζοντα. Μετά από κάποια ένσταση είχαμε κάποιο κώδικα διοντολογίας, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός. για όλες τις εκμεταλλεύσεις, τις γεωργικές. Όμως δεν εφαρμόστηκε. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η μόλυνση. Βλέπετε εδώ μία σπηλιά στο νότιο τμήμα της Μαγιόργα. Βλέπετε με το με κίτρινο το νερό αυτό που είναι γλυκό και καταλήγει σε μια φυσική λεκάνη με αυτό το γλυκό νερό. Όμως, έχουμε οργανικά στοιχεία και διάφορες βρωμιές που έχουν δημιουργήσει ένα ολόκληρο στρώμα εκεί. Να, βλέπετε εδώ πέρα σταλακτήτες που προέρχονται από, από τα ρηπογόνα στοιχεία, τα βρώμικα. και δίτες και, και πάνε σε αυτή την στόα και αντιμετωπίζουν αυτούς τους θαλακτήτες που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο βρωμιά. Να τα προβλήματα στις βαλερίδες. Και με τίποτα αυτό το, το, το σχέδιο της ε, λεκάνης δεν είναι λύση. Βλέπετε εδώ το διάγραμμα αυτό, πώς εξελίσσεται η αύξηση του, της περιεκτικότητας σε αρμυρό νερό. Εδώ τι γίνεται στην ίδια γιώτα, στο ίδιο πηγάδι. Βλέπετε την πρόοδο μέσα σε 10 χρόνια όπως το φαινομένο αυτό της του ε, θαλασσίου Και πάλι σκητά στον κύριο τρίζο μερα Όμως η γραμματεία μας δεν έχει λάβει κάποια στοιχεία, γιατί πρόκειται για πολύ πρόσφατη αναφορά. Άρα εξαρτώμεθα από τα όσα μας εξήγησατε προφορικά. Έχει το λόγο κύριε Ρωμένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην προηγούμενη αναφορά εκ νέου τίθενται ζητήματα τα οποία εντοπίζουμε ως δομικά προβλήματα στην Ισπανία όπως είναι η ανάγκη βελτίωσης του ελέγχου των αγιοτρήσεων, λήψη μέτρων για να πάψει η υπερεκμετάλλευση του δροφορορίζοντα. Επίσης εντοπίζουμε προβλήματα ρήπανσης του δροφορορίζοντα και ούτω καθεξής. Έγινε μια προκαταρκτική ανάλυση του δεύτερου υδρολογικού σχεδίου. Τα πορίσματα δείχνουν ότι επιμένουν πολλά από τα προβλήματα που εντοπίσαμε στο πρώτο υδρολογικό σχέδιο. Επομένως, ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νέο σχέδιο για τις Βαλεαρίδες και πρόσφατα ενημερώσαμε και το Εθνικό Συμβουλίο Ιδάτων. Στη γενική εισαγωγή μου είπα ότι με τον επαρκή έλεγχο των γεωτρήσεων ε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό γιατί επιλύονται κάποια ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόζονται οι γεωτρήσεις στου διαθέσιμου πόρου ε, για να επιτευχθούν και οι στόχοι τη καλή κατάσταση των υδάτων. Υπάρχει υπερεκμετάλλευση και βλέπουμε ότι είναι συγκεντρωμένη σε κάποια σημεία. Αυτό δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι ιωτρήσεις να μην ε, ξεπερνάνε το φυσικό όγκο του υδροφόρου ορίζοντα και να μπορεί να αναπληρωθεί ε, με φυσικό τρόπο ο υδροφόρος ορίζοντας. Επίσης, όπως είχα πει και στην πρώτη μου παρέμβαση, θα πρέπει να υπάρξει και κατά πολιτική τιμολόγηση για την ανάκτηση του περιβαλλοντικού κόστους ε, του νερού. και σε ό,τι αφορά τη χρήση πογείων υδάτων για υγειογικού σκοπού. Οι αρμόδιε αρχέ, λοιπόν λεκάνε απορρέσει, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα για να μπορούν να, να ασκούν τον απαιτούμενο έλεγχο και έτσι να εγγυηθούν και την ορθή διαχείριση και τον ορθό σχεδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αναφέρει αυτό το ζήτημα στις διμερείς επαφές που έχει αυτόν τον καιρό με τις Ισπανικές Αρχές. Ευχαριστώ. Thank you very much. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βαγίνα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω απλά να πω ότι πράγματι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Αναμένουμε την έκθεση. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές παρατυπίες και ατασταλίες. Άρα παραμένει ανοιχτή αναφορά και περιμένουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you very much and I see no... Ε, η πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανένα να γύρει ένσταση. Ακριβώς το ίδιο θα πρότεινα και εγώ. Πρόκειται για νέα αναφορά, άρα την διατηρούμε ανοιχτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε κάποια ανησυχία σχετικά με το υδρολογικό σχεδιασμό των Βαλεαρίδων νήσων. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρα μέτρα για να διατηρηθεί το οικοσύστημα. Αφήνουμε λοιπόν ανοιχτή την αναφορά και αναμένουμε περαιτέρω εξειδικευμένες. Α, με συγχωρείτε κυρία Ιούσο, δεν σας είχα δει. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Αυτό που ήθελα να ζητήσω είναι να ζητήσετε κι εσείς από πλευρά σας, από τους αναφέροντες, να ε, περιορίζονται στο θέμα. Η αναφορά ήταν ε, στην προκειμένη περίπτωση μια καταγγελία για το ότι δεν τηρούνταν οι, αρχή, οι όροι συγγνώμη, της δημόσιας συμμετοχής κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση δύο φορές ε, έγινε δημοσιοδεύει, ουσιαστικά ενημερώθηκε εκείνη η γνώμη. Δύο φορές. Εάν η αναφορά περιορίζεται σε αυτό το ζήτημα, ότι δεν έγινε δημόσια ενημέρωση, ζητώ από τους αναφέντες, όπως το ίδιο ισχύει και για, το, για την κοινοπραξία του Αλτο Γουαδιάνα. Μιλάνε για όλα τα έξω από το θέμα της αναφοράς. Και δράτω με τις ευκαιρίες αν μπορεί η Κομισιόν να μας πει, να μας δώσει τις εθνικές μελέτες για την εκτροπή στην περίπτωση του, ποταμού της Γρανάδας. Υπήρξε απόφαση και του ανώτατου δικαστηρίου. Τα στοιχεία αυτά είναι παλαιότερα, είναι καινούρια.